Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην 134η Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών. Καταρχήν, ως προς την ημερήσια διάταξη υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω αντίρρηση, οπότε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Μήπως υπάρχουν θέματα για τα πρακτικά της προηγούμενης μας Ολομέλειας. Δεν βλέπω αντιρρήσεις ούτε για τα πρακτικά, οπότε εγκρίνονται και αυτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα μέλη που ήταν παρόντα στην ε, τελετή εγγενείων του χώρου Παβέλ Ανταμόβιτς σήμερα το μεσημέρι, γιατί ο αγώνας του κατά της μισολαδοξίας και η προάσπιση των μειονοτήτων θα συνεχίσει να είναι πηγή έμπνευση για όλους μας. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω θερμότατα μια αντιπροσωπεία της τοπικής βουλής της Κάτω Αυστρίας ε, γιατί το γραφείο του στις Βρυξέλλες εορτάζει σήμερα τα 25 χρόνια αυτής της περιοχής ε, ε εκπροσώπησης μάλλον. Σας ε, καλωσορίζω θερμά. Επίσης, ε, μην ξεχνάτε τον οδηγό, το εργαλείο που έχουμε για, το ευρωπαϊκό, για τις ευρωεκλογές με πρακτικές πληροφορίες που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την σπουδαιότητα που έχουν οι ευρωεκλογέ. Επίσης, ένα φυλάδιο του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου για την κυβερνοασφάλεια είναι στη διάθεσή σας, στην είσοδο της αίθουσας. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές που καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε στα πλαίσια των ευρωεκλογών. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, Αγαπητή Δήμαρχε Μαντζινέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την σύνοδο της Ολομέλειάς μας με την παρουσίαση ενός νέου σχεδίου της Επιτροπής των Περιφερειών. Πρόκειται για την πρωτοβουλία Δήμη και Περιφέρειες για την ένταξη. Η πρωτοβουλία αυτή θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε τις τοπικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων άριθμα σχέδια έχουν δρομολογηθεί σε τοπικό επίπεδο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, στους μεγάλους δήμους, αλλά και στην Ήπεθρο που είναι πιο άρεο Και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή σε όλε τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ που βοηθούν του ερχόμενου να φτιάξουν μια καινούρια ζωή με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Γιατί είναι και αυτό το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να διστάζουμε, να αναδεικνύουμε τις θετικές εμπειρίες και τις επιτυχίες μας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης που πολύ, πολλές φορές τροφοδοτεί τη ρητορική του μίσους. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν υπέρ της ένταξης δεν εγκαινιάζεται μόνο από μας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως ε, στα πλαίσια της αστικής εταιρικής σχέσης για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών ε, που έγινε από την πόλη του Άμστερνταμ και τη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων. Επίσης, έχουμε τη βοήθεια των ε, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εδαφικών Ενώσεων, που είναι οι σύμμαχοι και εταίροι μας. Συνεργαζόμαστε και με άλλες οργανώσεις, όπως τον ΟΣΑ, την Τράπεζα Ανάπτυξης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Διεθνή ε, Καθολική Επιτροπή για τη Μετανάστευση στα πλαίσια των εκδηλώσεων που θα οργανώσουμε μέχρι τα τέλη του 2019. Βρισκόμαστε στην αρχή της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά ήδη 80 δήμοι και περιφέρειες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούμε. Από 17 χώρε μέλη προέρχονται αυτέ αυτές κοινότητε και περιφέρειες και στόχο μα είναι να καλύψουμε το σύνολο τη ε, επικράτηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στη συνεργασία μα ε, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ενισχυμένη χρηματοοικονομική υποστήριξη Ευρωπαϊκή Ένωση για του Δήμου και τι περιφέρειες που δίνουν μάχη υπέρ τη κοινωνική ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει τάχιστα να αποφανθεί για τι μελλοντικέ χρηματοδότησει στα πλαίσια και τη ε, εδαφική ανάπτυξη. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, Σήμερα αποδεικνύουμε ότι η επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών και προσφύγων είναι ταυτόχρονα και εφικτή και ευκταία και μάλιστα μερικές φορές έχει ήδη υλοποιηθεί. Η ένταξη είναι μια εποφελής για όλους επιχείρηση και για τις αξίες μας, για την αλληλεγγύη μας και για την εδαφική ανάπτυξη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας και πρώτα απ' όλα στον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξη και την παρουσία του και για την πολύ στενή συνεργασία που έχει με την Επιτροπή των Περιφερειών. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Merci, Monsieur Président. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μπορούσα να χάσω την ευκαιρία γιατί μπορώ να σας παρουσιάσω κάποια σχόλια, γιατί και εγώ ε, δεν τέλεσα δήμαρχο, όπω είπα στη δήμαρχο τη Αγκώνα. Γιατί από τη στιγμή που μια φορά είναι κανεί δήμαρχο, μένει για πάντα δήμαρχο. Κυρία Δήμαρχε τη Αγκώνα, χαίρομαι ιδιαίτερω που είστε παρούσα εδώ. Αγαπητά μέλη τη Επιτροπή των Περιφερειών, κυρίε και κύριοι, όπω είπα και προηγουμένω, χαίρομαι ιδιαίτερω για την παρουσία μου εδώ, για να συζητήσουμε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για το μέλλον και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε περισσότερες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Αν κάποιος με ρωτούσε ποια είναι η γνώμη μου και ποια κατά τη γνώμη μου είναι από τις βασικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες θα έλεγα η επιτυχής κοινωνική ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Δυστυχώς όμως αυτό το θέμα το αμελούμε πολύ συχνά. Το υποτιμούμε, το υποβαθμίζουμε, μερικές φορές και το παρανοούμε. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος. Εδώ δεν πρόκειται για κάποια ήπια μέτρα που απλώς καθησυχάζουν τη συνείδησή μας. Θέλουμε να προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια στους λεγόμενους αλλοδαπούς, όχι όμως στο εις των συμπολιτών μας. Το να καταστήσουμε εφικτή την ένταξη και επιτυχή ε, είναι θέμα που από τη πεπτουσία των οικονομιών και των κοινωνιών μα. Θα θέλαμε ένα τμήμα τη κοινωνία μα να μην συμμετέχει, να μην συμβάλλει, να μην συνεισφέρει στην κοινωνική ανάπτυξη. Θέλουμε ένα τμήμα τη κοινωνία μα να μην ομιλεί τη γλώσσα τη χώρα ή να μην μπορεί να έχει σχέσει με του υπόλοιπου πολίτε. Θέλουμε ένα τμήμα τη κοινωνία μα να νιώθει περιθωριοποιημένο, αποκλεισμένο, αλωτριωμένο ή ότι έχει υποστεί απόρριψη και ματέωση. Θέλουμε να διατρέξουμε τον κίνδυνο ένα τμήμα της κοινωνίας μας να στραφεί κατά της ίδιας της κοινωνίας. Κάθε άνθρωπος με κοινή λογική και κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το κοινό συμφέρον θα απαντούσε όχι φυσικά σε όλες τις προηγούμενες ερωτήσεις. Και να το πούμε με απλά λόγια. Το να επιτύχει η ένταξη έχει κρίσιμη σημασία για την συνοχή των κοινοτήτων μας και για την ευρωπαϊκή μας οικονομία. Ευτυχώς, αυτοί που εργάζονται ή απασχολούνται με το θέμα αυτό σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται την επιτακτική ανάγκη και τη σημασία που έχει η επένδυση σε αυτή την προτεραιότητα. Ως τοπικές και περιφερειακές αρχές γνωρίζετε κι εσείς ότι διαδραματίζεται σπουδαιότατο ρόλο στη διαδικασία αυτή γιατί δημιουργείται χώρους για ανταλλαγή απόψεων και για διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων εξασφαλίζοντας ένταξη κοινωνική και ενεργό συμμετοχή στο σύνολο της κοινωνίας. Και στηρίζεται αυτή την επαφή και το τέριασμα των μεταναστών με την τοπική αγορά εργασίας. Προωθείται την κοινωνική ένταξη μέσω παιδείας χωρίς αποκλεισμού και στέγη, στεγαστικής πολιτικής που δεν αποκλείει κανέναν. Επίσης συνεργάζεστε με τις ε, αντίστοιχες οργανώσεις επιτόπου και εντοπίζετε που υπάρχουν δυσφορίες ε, ή δυσχέρειες ή κάποια αναστάτωση. Γνωρίζω βέβαια ότι ουδή στην αίθουσα δεν είναι αφελής. Η ένταξη δεν είναι πάντα κάτι εύκολο. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, απαιτεί πολλές εργότες προσπάθειες και πολλές επενδύσεις από όλες τις πλευρές. Η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμπίπτει κυρίως ε, στην εντολή των εθνικών κυβερνήσεων. Αλλά και εσείς διαδραματίζετε ε, πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Και παρά τις προκλήσεις Έχουμε εκατοντάδε παραδείγματα τοπικών κοινοτήτων που έχουν καταφέρει να επιτύχουν την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων. Και εκεί η πολυμορφία είναι πλεονέκτημα, είναι ατού και όχι λόγος ανησυχίας. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα παραδείγματα να τα προβάλλουμε περισσότερο, να τα αναδείξουμε και να δώσουμε στους Δήμους και τις περιφέρειες περισσότερες ευκαιρίες για να παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους και να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Πιστεύω ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ε, για την ένταξη, η πρωτοβουλία δηλαδή που εγκαινιάζεται σήμερα κυρία Πρόεδρε, θα προσφέρει αυτό το χώρο και αυτές τις δυνατότητες. Πιστεύω ακράδαντα ότι έτσι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αφήγημα και μια πιο τεκμηριωμένη συζήτηση γύρω από την κοινωνική ένταξη και τη μετανάστευση. Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει και ενισχύει το έργο που έχουμε ήδη επιτελέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια προκειμένου να, εφαρμόσουμε έναν ε, καλό αμφίδρομο διάλογο μεταξύ των τοπικών περιφερειών και της κοινωνίας. Γιατί η ένταξη δεν είναι μόνο ε, λόγια, αλλά και έργα και μάλιστα συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Και γι' αυτό στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στις προσπάθειες εξασφάλισης κοινωνικής ένταξης και το κάνουμε αυτό με χρηματοδότηση, με κονδύλια από όλες τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές μας. Από το 2015 μέχρι το 2017 το Ταμείο Μετανάστευσης Ασύλου και Ένταξης συγχρηματοδότησε 4.800 μέτρα για να προαγάγουμε την ένταξη των ε, υπηκών τρίτων χωρών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να είμαι σαφής. Πρόκειται για χρηματοδότηση και υποστήριξη που πηγαίνει στους μετανάστες που ήρθαν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για κονδύλια που αφαιρούνται από τους Ευρωπαίους πολίτες ή που τα στερούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε ε, τις κοινωνίες μας και τις οικονομίες μας για να θάλουν, να ανθίσουν, θα πρέπει να στηρίξουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας μας. Έτσι θα καταστήσουμε την πολυμορφία ε, λειτουργική για όλους. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στην κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να είναι δύσκολη για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδιαίτερως για τις μικρότερες τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση για την ένταξη ε, προσπαθούμε να καταστεί πιο ε, προσβάσιμη για τις, τοπικέ για τις τοπικές αρχές στο μέλλον. Και γι' αυτό έχουμε αυξήσει και τα σχετικά κονδύλια. Κυρίες και κύριοι, ε, μια και έχουν μειωθεί τις σύλλου και παράτυπες αφήξεις σε επίπεδα πριν από την κρίση, έχουμε μια φόρα που έχουμε πάρει και μια όθηση για να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην κοινωνική ένταξη όσων έχουν ήδη έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω γιατί έχει νόημα κάτι τέτοιο, τι μετράει αυτό. Είναι αυτονόητο. Αλλά χρειαζόμαστε τη δική σα βοήθεια για να εξηγήσουμε το επιχείρημα αυτό στι εθνικέ κυβερνήσει. Θα πρέπει να υψώσετε τη φωνή σα και να περάσετε το μήνυμα για τα θέματα αυτά. Μην, Μην ξεχνάτε ότι ω δήμαρχοι και ω τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχετε πολύ ισχυρή πολιτική φωνή και γνωρίζετε πολύ καλύτερα την κατάσταση επιτόπου. Γιατί εσείς έχετε κάθε δικαίωμα αλλά και το κύρος ε, να μιλήσετε για τα θέματα αυτά και να απαιτήσετε υποστήριξη και μακροπρόθεσμες λύσεις. Γιατί αν δεν αλλάξουμε την οτροπία αλλά και το αφήγημά μας, η Ευρώπη κινδυνεύει να διαπράξει τα ίδια λάθη με τα σφάλματα των προηγούμενων δεκαετιών. Και εκείνα τα λάθη τα ένιωσαν όχι μόνο οι μετανάστες, αλλά τα ένιωσαν και οι δικές μας κοινωνίες. Η φωνή σας θα είναι σημαντική και στις επικείμενες ευρωεκλογέ. Η μετανάστευση και η κοινωνική ένταξη θα συζητηθούν ιδιαίτερο στην προεκλογική εκστρατεία και υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερους διχασμούς. Έχουμε λοιπόν κοινή ευθύνη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για μια πιο συνεκτική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος όλων των πολιτών μας και για αυτή την προσπάθεια η φωνή σας είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαντσινέλη, δήμαρχο της Ακόνα που πρόσφατα εξελέγει η δήμαρχος του κόσμου το 2018 και διαδέχτηκε τον Μπάσο Μέρτς. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπερτς για την πρόσκληση που μου απίθυνε για να συμμετάσχω στις εργασίες αυτής της Ολομελίας που για μένα είναι μεγάλη τιμή. Χαιρετίζω τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο. Συναντηθήκαμε και πριν την έναρξη των εργασιών. Χαιρετίζω όλη τη συνέλευση. Κυρίως θέλω να απευθύνω χαιρετισμό προς τον συνάδελφο Σόμερς που ήταν ο δήμαρχος του κόσμου το 2016, World Mayor ε, και ήταν ε, χαρά μου να το συναντήσω προσωπικά για να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά για τη μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι περίπλοκο το θέμα ε, και έχει διάφορε πτυχέ. Ανάλογα από την οπτική γωνία, θα ήθελα να αναφέρω δύο πτυχέ. Η πρώτη αφορά την ένταξη των ανθρώπων, των αλλοδαπών που δίνουν, ζουν παράτυπα στην πόλη μου. Το δεύτερο θέμα είναι διαφορετικό ε, και αφορά τι ανεξέλεκτε ροέ μεταναστών που έρχονται κυρίω σε αυτή την περίοδο από την Αφρική και που αυξάνονται εκθετικά τα επόμενα, θα αυξηθούν εκθετικά τα επόμενα χρόνια και ίσως αφορά αυτό και την πόλη μου την Αγκώνα, υπέροχη πόλη στην Αδριατική, ε, έχει μια χεσόνησο ε, ε, και είναι μια πόλη που κάνει την ταυτότητά της, στη θάλασσα ταυτότητά της. Είναι ένα θέαμα καθημερινά, είναι σημαντικό λιμάνι διεθνές, οι ηγίτες της διασυνδέσεις ε, με την Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη. Έχει, έχουμε εκεί παραγωγή ναυπήγηση σκαφών κρουαζιέρας και τα καλύτερα γιότ παράγονται εκεί. Έχουμε πάρα πολύ μακρι, χρόνια ύπαρξη σαν ζωή και αναγέννηση πέρας από από εμά προφανώς και ε, ε, είχαμε και τους πρώτους πίνακες του Τιτσιάνο και τους τελευταίους πίνακες αυτού ε, έχουμε του πρώτου πληθυσμού που ήρθαν από την Αλοδαπή. 30 μέχρι 40% έχουμε Αλοδαπού στην πόλη. Ε, πάνω από 100 διαφορετικέ εθνότητε έχουμε. Δεν έχουμε ακραίες, ε, ακραία προβλήματα όπω έχουν οι μεγάλε Μητροπόλει, αλλά να πούμε ότι η συμβίωση είναι κάτι εύκολο είναι να πούμε κάτι που δεν ισχύει. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίζεται καθημερινά, έλεγε πριν ο Επίτροπο, ο κ. Αβραμόπουλο. Είναι ένα πρόβλημα να αντιμετωπίζεται καθημερινά. Δεν πρέπει να ρίχνουμε οξυγόνο στη φωτιά όπως κάνουν οι διάφοροι ακραίοι στην ε, Ευρώπη αλλά ούτε να λαχιστοποιούμε και να αρνούμεθα την ύπαρξη του προβλήματος. Η ένταξη δεν είναι μόνο κάτι σωστό και δίκαιο αλλά είναι και βολικό για όλους. Αλλά είναι με μακρά και κοπιαστική διαδικασία και δεν είναι κάτι αυτόματο. Απαιτεί χρήματα, πόρους, πολιτικές συνεχείς από τη... στο σχολεία πρέπει να ξεκινά σε εμά, ήδη ε, στο δημοτικό, να ενημερωθούν, να μάθουν τα παιδιά πώ να έχουν και επαφή, να, ανήκουν, να έχουμε αγωγή του πολίτη. Ε, πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι μόνο θέμα που αφορούν του διδασκάλου. Ε, χρειάζονται υποστήριξη διδασκαλή και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σαν κοινότητε έχουμε πολλές πολλά προγράμματα. Έχουμε εθνικά προγράμματα, συνδέσει με διάφορου φορεί για μαθήματα ένταξη Χρησιμοποιούμε και ένα άλλο σημαντικό κανάλι για να διευκολύνουμε την ένταξη των οικογενειών που ζουν σε εμά ε, με ε, άδεια διαμονής και εργασίας. Ποιος διάβλος είναι αυτός, οι γυναίκες, οι μητέρες. Είναι αυτές που συμμετέχουν περισσότερο στα μαθήματα γλωσσών, βασικό εργαλείο για την ένταξη και για την αγωγή των πολιτών. Όλα αυτά Μα δείχνουν ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση εάν η μετανάστευση είναι διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη εντός των ορίων τη νομιμότητα και της ασφάλειας. Αλλά δεν ισχύουν τα ίδια για την ανεξέλεκτη και την παράτυπη μετανάστευση. Οι μεταναστευτικέ ροέ τείνουν να αυξάνονται, κυρίω από την Αφρική και από αυτέ τι περιοχέ όπου οι αλλαγέ του κλίματο καθιστούν ε, το βίο-βίο του σε μεγάλε περιοχέ όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν μπορεί ε, να υποδεχθεί όλου η Ευρώπη. ή Θα διαλυθούν οι πόλει μα. Ανοιχτέ πόρτε ναι, αλλά ανοιχτέ πόρτε δεν μπορεί να συμβαίνει σύνορα ανοιχτά. Να σημαίνει κάτι τέτοιο. Ανοιχτά λιμάνια και ανοιχτέ πόρτε σημαίνει να σώζουμε τις ζωές, να σώζουμε από την απελπισία τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα. Ένα, ε, λοιπόν, ένα κράτος πρέπει να τους διασώζει αυτούς αν δεν θέλει να χαθεί η αξιοπρέπειά της. Αλλά πρέπει να ελέγχονται οι ροές και θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πολιτική για την Αφρική που θα βελτιώνει τις συνθήκες ζωής αυτών των πληθυσμών και που εκεί πρέπει να πρωταγωνιστεί η Ευρώπη. Το θέμα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό και σήμερα δεν είναι κάτι τέτοιο. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την ευθύνη να αναλάβει ένα τμήμα των ανθρώπων που καταφθάνουν ε, και που θα γίνουν δεκτά. Αυτός που δεν θέλει να το κάνει δεν μπορεί να νίκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κανείς να είναι εθνικιστής αυτές τις μέρες και να εμποδίσουμε τους μετανάστες να μπουν σε μια χώρα και να μην είμαστε όταν μπαίνουν τα κεφάλαια, να μην δείχνουμε προστατευτισμό, οι επενδύσει των επιχειρήσεων και ίσω από άλλε χώρε τη Ένωση, που μετεκαθίστανται σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχει χαμηλότερο κόστος εργασίας και να το πούμε ειλικρινά όπου τα δικαιώματα των εργαζομένων πολύ συχνά είναι μικρότερα. Η Ευρώπη πολύ συχνά υποστηρίζει και αυτές τις πρωτοβουλίες σε χώρες που μετά με ανεύθυνο τρόπο παραμένουν ε, με κοφά όταν αφορά τα για υποδοχή των μεταναστών. Αυτή, αυτή η διαφορά οδηγεί σε μια, ένα κίνδυνο σώριξη της Ευρώπης. Θα πρέπει να είναι γίνει ισότιμη η Ευρώπη για όλα τα θέματα, μετανάστευση, δικαιώματα εργαζομένων σε όλους τους τομείς. Μόνο έτσι θα μπορούμε να επιλύσουμε και στην τρίτη χιλιετία ε, ε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ε, που αντιμετωπίζουμε και να τηρήσουμε τι αξίε μα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπω έλεγε και ο επίτροπο στην αρχική του παρέμβαση, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά ούτω ώστε να εισακουστούν και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Χρειάζεται όσον αφορά το θέμα της ένταξης και για να ανταποκριθούμε στις εσφαλμένες πολιτικές εκείνων που τροφοδοτούν τη μυσαλλοδοξία, που τροφοδοτούν την αντιπαράθεση, των πόλεμο μεταξύ φτωχών για να ανταποκριθεί σε εσφαλμένες πολιτικές θα πρέπει όσον αφορά την ένταξη να έχουμε λιγότερη ρητορική και περισσότερη δράση, περισσότερους πόρους και περισσότερες πολιτικές οργανωμένες χρονικά αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι και θα είναι το πρόβλημα του αιώνα που έχουμε μπροστά Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντσινέλη. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους και στους εκπροσώπους των τεσσάρων ε, οργανώσεων που είναι μαζί μας. ΑΕΡΕ, ΣΕΜΕΡ, ΣΕΠΕΑΡΕΜ και EuroCities. Ένα, ένα λεπτό παρακαλώ καθένα. Ο κύριο Επίτροπο πρέπει να φύγει στι θέσει, αλλά θα ήθελα να έχει δυνατότητα να, να έχει δυνατότητα να απαντήσει. Μόλι θα πάρει το λόγο και ο κύριο Ματιού Λεκλέρ που θα εκπροσωπεί το EuroCities, η πρόεδρο τη Επιτροπή μα ΣΥΒΕΞ, κυρία Μπάρμπαρα Ντούρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ήδη στο παρελθόν επανειλημμένα είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με το σημαντικό θέμα ένταξη των προσφύγων και πόσο απόλυτα αναγκαίο είναι να υπάρχει στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της Ένωσης για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα κάναμε ένα σημαντικό ε, συμβολικό βήμα με την έγκριση αυτής της έκθεσης στις ε, πόλεις και τα χωριά μας δεν έχουμε καμία εναλλακτική λύση από την ένταξη. Αλλά, αν είμαστε ειλικρινεί, δεν είναι μόνο λύση ενό προβλήματος αυτή η ένταξη, αλλά είναι βάση και για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας για το μέλλον μας. Η ένταξη δεν αφορά μόνο τους ε, νέο αφικνόμενους, αφορά, αφορά τις κοινότητες ε, συνολικά γιατί αλλιώς διευκολύνουμε αυτούς που θέλουν να εντείνουν τις κοινωνικές διαφορές λέγοντας ότι τα λεφτά τα παίρνουν οι μετανάστες και εμείς οι αποκλεισμένοι όχι. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τον τρόπο ε, της ένταξης, για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων σε όλες τις περιοχές της Ένωσης. Η Ένωση έχει πολλές επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα, όπως ξέρετε, με από το Αμβούργο. Μια πόλη που ούτε μικρή ούτε ιδιαίτερα φτωχή είναι. Αλλά ακριβώς σε μια πόλη όπως το Αμβούργο βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις ε, των κοινωνικών διχονιών είναι σημαντικός κίνδυνος για την κοινωνία μας. Στην ε, πόλη μου έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες αλλά και έντονη συζήτηση με τους εταίρους μας και στην Ένωση και ευρύτερα από όπου επωφεληθήκαμε. Έτσι βλέπουμε σε τι επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και με τι τρόπο. Μαθαίνουμε εμένα από τους δε. Ελπίζω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία αυτή πόλεις και περιφέρειες για την ένταξη θα είναι ένα περαιτέρω βήμα και θα στηριχθεί και από την ε, τωρινή και από την μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος, ο κύριος Μάγνους Μπέρτσον, Πρόεδρος της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης. Κυρίε και κύριοι, η περιφέρεια των, ε, συγγνώμη, η συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης ε, εκτιμά ιδιαίτερα αυτή τη συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών που θεωρώ πως είναι ένας από τους κύριους εταίρους μας στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη είσοδο μεταναστών και προσφύγων. Μπορεί να έχουν μειωθεί αυτές οι ροές, αλλά παραμένουν οι πιέσεις. Η αύξηση των αφήξεων στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο είχε ω συνέπεια η στήριξη των ε, κοινοτήτων και πόλεων που αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό να είναι προτεραιότητα για την Ένωση. Πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης. Έχουμε τρόπο για να βοηθήσουμε την ένταξη μεταναστών και προσφύγων να συμβάλλουμε στην κοινωνική, οικονομική και ε, στην εκμάθηση των ε, πολιτικών μας αρετών. Γιατί η Ευρώπη θα ωφεληθεί από αυτή την ε, πολυφωνία. Και αυτό είναι προτεραιότητα για την πολιτική μας εργασία. Δημιουργήσαμε μια ειδική ομάδα, Task Force, μεταξύ Καταλωνίας, συγγνώμη που, της οποίας προεδρεύει η Καταλωνία, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να μάθουμε μένα από τους δε. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα AMID για τους μετανάστες ε, με αναπηρίες. Αν η Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις δεν δημιουργήσουν ένα επαρκέ σύστημα διακυβέρνησης, εάν δεν ενισχύσουν την οικονομική στήριξη προς τις περιφέρειες για να παίξουν τον θεμελιώδη ρόλο τους στην ένταξη των αφιγνουμένων και να δημιουργήσουν κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, θα είναι δύσκολο η Ευρώπη να επιτύχει τη διαχείριση της μετανάστευσης και να ωφεληθεί από την ε, πολυμορφία των κοινοτήτων της και να δημιουργήσει κοινωνίες με συνοχή. Γι' αυτό η οργάνωσή μου καλωσορίζει αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιφερειών θα προσφέρει στις κοινωνίες και στις πόλεις πλατφόρμες για να συνεργαστούμε για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ελένη Λουκαίδου από την Επιτροπή των Περιφερειών. <coughs> Κύριε Επίτρεπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα πρέπει να πω ότι η Κύπρος τον τελευταίο καιρό κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αναλογία πληθυσμού στην άφηξη παράνομων μεταναστών ο δήμος λευκοσίας στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για κοινωνική στήριξη και ευαισθητοποίηση προχώρησε στην ίδρυση ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού του πολυδύναμου δημοτικού κέντρου λευκοσίας βασική στόχη του οποίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου. η αφοσίωση και η δέσμευση της λευκοσίας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρει κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες είναι ζωτική σημασίας. Μέσω του πολυδύναμου υλοποιούνται προγράμματα και προσφέρονται ποιοτικέ υπηρεσίες φροντίδας, απασχόλησης, ψυχοκοινωνική στήριξης, διαβίου μάθηση, επαγγελματική και κοινωνικής επανένταξης σε ευάλωτε ομάδες και σε μετανάστες. Πιστεύουμε ότι με τη σωστή στήριξη οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, γίνονται πηγή δημιουργίας και εμπλουτίζουν την τοπική ζωή. Η Λευκοσία, μια πόλη που ανέκαθεν υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών, θα παραμείνει μια ανοιχτή πόλη. Για 8η συνεχή περίοδο υλοποιούμε το πρόγραμμα Νέοι δρόμοι για την ένταξη με συγχρηματοδότηση 90% από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δράσεις του δήμου περιλαμβάνουν προγράμματα κοινωνικής στήριξης σε μετανάστες και λειτουργία κέντρου ενημέρωσης και υποστήριξης. επίσης προγράμματα δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό και την κοινωνία της κύπρου με πρωτοποριακά εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας για παιδιά και τη δικτύωση των μεταναστευτικών οργανώσεων με τις τοπικές αρχές για τη συστηματοποίηση δράσεων ένταξης. Παρέχεται επίσης κοινωνική στήριξη και οργανώνονται πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες συγχρονισμού των μεταναστών και του ντόπιου πληθυσμού, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με στόχο τη διατήρηση των πολιτισμικών στοιχείων της καταγωγής τους καθώς και εργαστήρια σεμινάρια σε ενήλικες. Αυτά εν συντομία. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γουί Μπετανκούρ εκ μέρους της διάσκεψης των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή που το θέμα της μετανάστευσης έχει γίνει πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και για, την ε, Ευρω... και για τον κόσμο. Εμείς ε, που εκπροσωπούμε εκατοντάδες ε, περάκτες περιφέρειες έχουμε ιδιαίτερη επίγνωση του προβλήματος. Γι' αυτό από το 2015 ξεκινήσαμε να εντρυφούμε στο θέμα της μετανάστευσης και έχουμε πρωτοβουλία σε πολλές μεσογειακές περιφέρειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την κοινωνική ένταξη των μεταναστών οργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συστήνεται και μία ομάδα εργασίας που φέρνει σε επαφή πολλές χώρες ε, προέλευσης, ε, διέλευσης ε, και προορισμό. Επίση, έχουμε εκπρόσωπο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την ομάδα αυτή εργασία έχουμε συγκεκριμένε προτάσει για τον ρόλο των ιδιαίτερα των παράκτων περιφερειών. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το δυναμικό των περιφερειών, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση της ένταξης. Θα βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη να το επιτύχουν στην... Για τη μεταναστευτική πολιτική έχουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Γι' αυτό ζητούμε πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση και κονδύλια για τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά δεν αρκούν η παρούσα κατάσταση σε ό,τι αφορά τι μεταναστευτικέ ροές αλλά και η γεωπολιτική κατάσταση σε πολλέ γειτονικέ χώρες της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας ε, να ενισχύσουμε τις αμοιβέ μας ικανότητες γι' αυτό και η διάσκεψη Παράκτητων περιφερειών θέλει να συνεργαστεί με την Επιτροπή των Περιφερειών και να συμβάλλει με το έργο τη και τι πρόσφατε πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε για τι προοπτικέ στις περιφέρειες αυτές να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικέ για το μέλλον και στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και να κάνουμε μια καλή χαρτογράφηση ε, των ικανότητων που χρειαζόμαστε και, για την καλύτερη διακυβέρνηση ε, με εκμεταλλευόμενη τις εμπειρίες των περιφερειών. Ευχαριστώ το λόγο ο κύριος Μπάρτ Σόμερς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι, μάδα ομάδα μου χαίρεται πάρα πολύ για την πρωτοβουλία των πόλων και των περιφερειών, για την ένταξη η σημερινή πραγματικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία καταστάσεων και πρέπει να το δεχτούμε. Η μετανάστευση συχνά θεωρείται κάτι αρνητικό και μπορεί να αποτελέσει υποστηθέμενη αξία. Θα πρέπει να κάνουμε πράγματα και να μάθουμε εμένα από τους ΔΕ. Ένα δίκτυο από πόλεις με καλές πρακτικές μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε βεβαίω, να δώσουμε στους μετανάστες τις δεξιότητε, να συμμετάσχουν ενεργά στις κοινωνίες μα. Πρέπει να, σε θέση, να είναι σε θέση να μάθουν τη γλώσσα, αλλιώς απομονώνονται. Πρέπει να έχουν ευκαιρίες να βρουν δουλειά πρέπει να μπορούν να ανήκουν στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, επίση, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε να καταπολεμήσουμε την απομόνωση τη πόλη μα. Λέμε ότι η ποικιλομορφία είναι προστιθέμενη αξία. Στην πραγματικότητα, πολύ συχνά ζούμε σε ένα αρχιπέλαγο πολυεθνικών ε, νησιών. Και η ποικιλομορφία μπορεί να είναι προστιθέμενη αξία αν είναι ένα κομμάτι τη καθημερινή σου ζωή, αν συναντά ανθρώπου, εάν συγχρονίζεσαι με ανθρώπου με διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό πρέπει να αφήσουμε πίσω μα είναι ομαδική νοοτροπία, κοινοτική νοοτροπία. Αν δούμε στι πόλει, όλοι έχουμε την τάση να διαιρούμε σε ομάδε, σε κοινότητε τη πόλη. Δίνουμε μία ταυτότητα στου ανθρώπου, βάζουμε σε μία ταυτότητα, του βάζουμε σε κουτιά και βάζουμε ετικέτα στα κουτιά. Καμιά φορά θεωρούμε ότι είναι θύματα οι άνθρωποι διακρίσεως. Θεωρούμε ότι καμιά φορά καταχρώνται του κοινωνικού συστήματος. Πολύ συχνά όμως εθελοτυφλούμε όσον αφορά τα θετικά πρότυπα που υπάρχουν. Υπάρχουν κατάδε σε κάθε πόλη που να δώσουν κίνητρα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, να δώσουν κίνητρα να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις για να κάνουμε τη διαφορά στην κοινωνία μας ούτω ώστε το πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε γενικού τίτλου στου ανθρώπου. Πρέπει να δεχτούμε ότι ταυτόχρονα οι άνθρωποι έχουν διαφορετικέ ταυτότητε και αυτό είναι προστιθέμενη αξία. Τέλο, να πω ότι πρέπει η κοινωνία να βασίζεται σε κοινέ αξίε. Πρέπει να υπερασπιστούμε τι αξίε. Μία από τι βασικέ αξίε όμω τη κοινωνία μα είναι η καταπολέμηση του ρατσισμού και τη διάκριση. Και πολύ συχνά από τη λαϊκιστική πλευρά ξεχνούμε ότι ότι όλα αυτά ανήκουν στο δυτικό μας πολιτισμό. Όλοι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για τους εαυτούς τους και για την κοινότητα στην οποία ζουν. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή, Πιέτρο Πούτσιο για το Συμβούλιο των, Κοινο... των Περιφερειών της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί Δήμαρχοι, και εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκησης είναι τιμή για μένα να απευθύνω σε εσά και να μιλήσω σαν εκπρόσωπο του Συμβουλίου των Κοινοτήτων και των Περιφερειών της Ευρώπης όσον αφορά την πρωτοβουλία πόλη και περιφέρειες για την ένταξη. Το Συμβούλιο των Κοινοτήτων και των Περιφερειών της Ευρώπης αντιπροσωπεύει πάνω από 100.000 εκπροσώπου τοπική αυτοδιοίκησης, φορεί σε 55, από 55 εθνικού συνδέσμου, τα τελευταία χρόνια εργάστηκε για τη βελτίωση τη ένταξη των μεταναστών, των ετούντων άσυλο και των προσφύγων και για να δημιουργηθούν πόλει και περιφέρειες που καλύπτουν περισσότερου. Ε, κάναμε διάφορα ψηφίσματα στην Επιτροπή των Περιφερειών και τοποθετηθήκαμε βάσει αρχών που θα πρέπει να κατευθύνουν τι απαντήσεις Ευρώπη, ανθρωπιστικέ απαντήσει στην διαθροτική πρόκληση τη ε, μετανάστευση, από πλευρά ε, τοπική και περιφερειακή, διότι στο Τέλος, η ένταξη σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει πιο συνεκτικές κοινωνίες, Μόνο όμω μπορούμε να το πετύχουμε αυτό αν έχουμε πιο συνεχτικέ πόλει. Αυτό το στόχο είχαμε. Να βελτιώσουμε την άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ενισχύσουμε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Ε, για να προωθήσουμε πιο ευέλικτη πρόσβαση στη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να βελτιώσουμε την πρόσβαση υπηρεσίε για του πρόσφυγε και του μετανάστε σε επίπεδο τοπικό μέσω τη δημιουργία ε, ενία θηρίδα. Όλη αυτή η δουλειά μαζί με εκείνο των δικτύων τη Επιτροπή των Περιφερειών είναι κάτι που ενισχύει τη βαθιά δικιά μα σύμφωνα με την οποία αυτέ οι πρωτοβουλίε είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου ή προ τη σωστή κατεύθυνση για να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτική και να βελτιώσουμε την ανταλλαγή γνώσεων ε, εν ώψη των ευρωεκλογών των επικειμένων και σε μια στιγμή όπου κάποια κράτη-μέλη και κάποιοι πολιτικοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη μετανάστευση σαν ένα μέσο για να οδηγήσουν αντιπαράθεση και να μειώσουν τις κοινέ μα αξίε, οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι στην πρώτη γραμμή για την υποδοχή των προσφύγων και την παροχή υπηρεσιών στου πολίτε τρίτων χωρών. Ε, εμείς συμμετείχαμε στην σύμπραξη για την ένταξη των προσφύγων μεταναστών στο θεματολόγιο τεστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν μια πλατφόρμα επιτυχής για να προωθήσουμε την αρχή της σύμπραξης, της συνεργασίας και να έχουμε ε, επιρροή όσον αφορά την νομοθεσία της πολιτικές κάνοντας και προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Πέρασε ο χρόνος αγορεσή σας. Θα πρέπει να έχετε Είχατε δύο λεπτά και έχετε ξεπεράσει κατά 30 δευτερόλεπτα. Θα μα εγκαταλείψει ο κύριο Επίτροπο τώρα, διότι στι 4 ε, έχει σημαντική συνεδρίαση. Θα του δώσω συντομία το λόγο για να απαντήσει σε εκείνου που ήδη του μπόρεσαν να λάβουν το λόγο. Σα ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος ε, Σόμερ. Το θέμα είναι αξιών είναι θέμα αξιών και αρχών, γιατί οι δημοκρατίες βασίζονται σε αυτές τις αξίες. Και ακριβώς η κρίση του μεταναστευτικού έθεσε εν κινδύνο αυτές τις αρχές. Ορισμένοι τις αμφισβητούν, τις αξίες και τις αρχές αυτές. Άρα πρέπει να δώσουμε μια πολύ σαφή απάντηση. Και δεν διστάζω να πω ότι από τότε που ε, ανάλαβα τα καθήκοντά μου αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Και τώρα, επειδή επίκυνται ευρωεκλογές, απειλούμεθα όλοι από την άνοδο της, ε, του λαϊκισμού καθώ και του εθνικισμού. Όλοι αυτοί θέλουν να υπονομεύσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οπότε όλοι, είτε η Επιτροπή είτε τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό όραμα. Ε, η κυρία Ντούντεν μου έκανε μια ερώτηση. Να σας δώσω περισσότερες προφορίες για το τι κάνουμε ως Επιτροπή. Από την αρχή η Επιτροπή στήριξε ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Περιφερειών. Βοηθήκαμε, βοηθήσαμε, στηρίξαμε, κινητοποίησαμε τις τοπικές αρχές για να προωθήσουμε την ένταξη. Η Επιτροπή έχει συντονίσει στην προσπάθεια αυτή το, την εταιρική σχέση για το αστικό θεματολόγιο, για τα θέματα ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην πόλη του Άμστερνταμ και έχει στηρίξει απευθείας τις πόλεις και τις περιφέρειες μέσω χρηματοδότηση από το ΑΜΙΦ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεργαστεί για το θέμα της ένταξης με τη δική σας Επιτροπή. Οπότε, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας που μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον για το θέμα αυτό. Τώρα, οι δράσεις της Ένωσης για την ένταξη στις πόλεις. Γιατί θέσατε το θέμα αυτό κύριε Μπέλτσα. Ένα απτό παράδειγμα του διαλόγου που έχουμε δημιουργήσει είναι η εταιρική σχέση για την ένταξη των ε, προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος για την αστική αναγέννηση. Έτσι συνεργάζονται όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό με τους ίδιους τους μετανάστες. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση πριν από μια πενταετία, αυτή η συνεργασία τότε που ξεκίνησε, τότε δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία. Τώρα γίνει πραγματικότητα. Σα στηρίζουμε όλου απευθεία. Οικονομικά, λειτουργικά και συγκεκριμένα. Η Επιτροπή Περιφερειών είναι πολύ ενεργό τμήμα αυτής της συνεργασίας και ευχαριστώ τον Πρόεδρό σας και σε όλους και όλους εσάς ευχαριστώ η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της ε, συνεργασίας για παράδειγμα θα έχει ως αποτέλεσμα τον προσεχή Μάιο την δεύτερη εκδήλωση της Αστικής Ακαδημίας για την ε, ένταξη και ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την κατάρτιση των τοπικών αρχών και οργανισμών που ασχολούνται με την κατάρτιση ακριβώς των μεταναστών. Τώρα για τη χρηματοδότηση. Θα ξέρετε, προτείνουμε ουσιώδη αύξηση της ε, ενωσιακής χρηματοδότησης για τη μετανάστευση και τα σύνορα, επί τρία, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο θα έχουν ως θεματική προτεραιότητα τη μετανάστευση. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά των ταμείων αυτών για τη μετανάστευση όπου υπάρχει ανάγκη επιτόπου οι τοπικές αρχές σε στενό συντονισμό με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των ταμείων αυτών θα πρέπει λοιπόν να δράσουν για να εφαρμόσουν τα εθνικά προγράμματα ένταξης. Τώρα, στην κυρία Λουκαίδου θα απαντήσω ελληνικά. Λουκαίδη πρέπει να σας πω ότι όπως είναι γνωστόν εξάλλου παρακολουθώ το τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Πρόσφατα ήμουν και στην Κύπρο ενημερώθηκα και από τις εθνικές αρχές αλλά και από τις τοπικές αρχές και θα ήθελα πραγματικά να εξάρω την πόλη της Λευκοσίας για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Είναι ένα καλό παράδειγμα μιας μικρής πρωτεύουσα με ανοιχτές τις πόρτες που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι και το πνεύμα που κυριαρχεί στην Επιτροπή των Περιφερειών. θα ήθελα να πω και κάτι απλό. Αν οι εθνικές κυβερνήσεις άκουγαν περισσότερο τις τοπικές αρχές θα κυβερνούσαν καλύτερα και το κυριότερο θα κυβερνούσαν με αρχές και αξίες. Έχετε την απέριστη στήριξή μας σε αυτό που ήδη στέλνει στην Κύπρο γνωρίζοντας ότι η Κύπρος αυτό τον καιρό τελεί κάτω από μεγάλη πίεση και επειδή δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον και επειδή η Κύπρος είναι στις παρυφές ενός μεγάλου τόξου αστάθειας θέλω να ξέρετε και να μετεβάσετε και στι τοπικέ και στις ελληνικέ αρχές την αμέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και της Ευρώπης. Τελευταία θα ήθελα να αναφερθώ στο, στα MFF. On MFF uh, ε, synergies... Για τις συνέργειες του πολιτού δημοσιογραφικού πλαισίου για την ένταξη. Είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρχει συμπληρωματικότητα με τα άλλα ταμεία. Direction. synergies with the structural funds migration. Οι προτεραιότητέ μα είναι ακριβώ η ασφάλεια και η ένταξη. Όλα αυτά καλύπτονται από τον κανονισμό των διευθυντικών ταμείων. Για παράδειγμα, τα μέτρα ένταξη του κοινωνικού ταμείου, του δείκτε και φυσικά μέσω του κανονισμού για τι κοινέ διατάξει. Για παράδειγμα, αν θέλετε να σημειώσετε, η Επιτροπή προτείνει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ένα συνολικό, μια συνολική χρηματοδότηση πάνω από 100 δις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για την ένταξη, για κοινωνικές ενέργειες, για ένταξη στην κοινωνική αγορά και τη βοήθεια ε, σε ευάλωτες ομάδες ε, όπως συμπεριλαμβάνονται και οι πρόσφυγες. Αλλά επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα να χάσω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σα και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μεγάλη στήριξη <clears throat> που μας δίνει από την αρχή η Επιτροπή σα, ούτω ώστε να μπορούμε σήμερα να πούμε ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο από την εποχή τη έναρξη της κρίσης ουσιώδη πρόοδο και ελπίζω ότι στο μέλλον η Ευρώπη θα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Αλλά να μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το πρώτο επίπεδο οποιασδήποτε διοίκηση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα είναι <clears throat> τοπικέ αρχέ και περιφερειακές αρχές. Επαναλαμβάνω, έχετε την πλήρη στήριξή μα και συγκεκριμένα και οικονομικά και λειτουργικά. Σε ευχαριστώ πολύ για την θαυμάσια αυτή συνεργασία που είμαι πεπισμένο ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Θα δώσω το λόγο στο μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, τον κύριο Κάρλ Βαν Λόου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα του Επιτρόπου, αλλά είναι κρίμα πραγματικά που έφυγε στα μισά της συζήτησης. Πάντως, ήδη ακούσαμε πολλές φορές ότι η ένταξη δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες ε, για, τις, το, για τους Δήμους και τις περιφέρειες και αγγίζει και την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα θετικό αφήγημα γύρω από τη μετανάστευση και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι ναυηχθέντες ε, να, να παρακολουθούν μαθήματα αγωγής του πολίτη για να μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στην τοπική κοινωνία. Δεν μπορούν να είναι ε, παόριστον νέο αφιχθέντες, νέο εισερχόμενοι, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν αναπόσπαστα μέλη της κοινωνίας που τους ε, υποδέχθηκε. Και στην Φλάδρα έχουμε εδώ και χρόνια τέτοια μαθήματα αγωγής του πολίτη που εδράζονται σε τρεις πυλώνες. Καταρχήν εκμάθηση της γλώσσας. Είναι απαραίτητη εκμάθηση της τοπικής, της εθνικής γλώσσας. Αυτό διευκολύνει τις διαπροσωπικές επαφές με τους γείτονες, τις ε, αρχές, το δημόσιο, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο και ευνοεί και τις, τις εργασιακές προοπτικές. Επίσης, ε, καλύτερη κοινωνική ένταξη. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι μετανάστες σε τι κοινωνία ε, εισήλθαν. Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν αυτή την κοινωνία, οι αρχές, οι αξίες, τι δικαιώματα και τι υποχρεώσει έχουν ω μέλη αυτής της κοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και της τοπικής αγοράς ε, επαγγελματικές για να εξασφαλίσουμε ένα είδος επαγγελματικού προσανατολισμού στους ε, μετανάστες και πρόσφυγες. Και φυσικά κάποιος, ε, κάθε ένας ερχόμενος έχει ατομικές ανάγκες. Θα πρέπει περιπτωσιολογικά και μεμονωμένα να εξετάσουμε τις ανάγκες του καθενός και επίσης ε, να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του καθενός και τις κοινωνικές ανάγκες και να τις συντεριάξουμε καλύτερα. Χρειάζεται να αφιερώσουμε πολλές προσπάθειες στην προσέγγιση αυτή και ελπίζω με την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Δήμαρχο τη Γάλλη, ο κ. Ματία Δεκλέρκ, εκ μέρου των EuroCities, των Ευρωπαϊκών Πόλεων. Εκ μέρου των Ευρωπαϊκών Πόλεων του EuroCities θα ήθελα να σα ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση που μα κάνατε και τα δύο λεπτά που μα δίνετε για να συζητήσουμε ε, εξ των 140 εκατομμυρίων πολιτών που εκπροσωπεί το δίκτυό μα το EuroCities. Θα ήθελα να κάνω κάποιε δηλώσει. Τα τελευταία χρόνια η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η ένταξη στην αγορά εργασία των μεταναστών και προσφύγων. Αλλά η μοναδική επικέντρωση στην οικονομική ένταξη και στην αγορά εργασία δεν αρκεί. Η κοινωνική ένταξη, η στέγη και η πρόσβαση στην παιδεία είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες και προκλήσεις της ένταξης που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Δεύτερον, οι πόλεις, οι δήμοι έχουν καινοτόμες και επιτυχείς ε, πρακτικές για να ε, υλοποιήσουν αυτή την ε, ένταξη. Έχουν ειδικές ομάδες για να λειτουργήσει η η ένταξη από κάθε άποψη. Για παράδειγμα η πόλη της Γάνδης έχει συστήσει μια ομάδα κρούσης ε, για τους πρόσφυγες. Ε, εξασφαλίζεται συνεργασία μεταξύ του δημοσίου, της κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των πολιτών για να ε, στεφθεί με επιτυχία η κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Επίσης, οι πόλεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να καταρρύψουν το αρνητικό αφήγημα γύρω από τους μετανάστες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα στις πόλεις όλοι οι πολίτες να αναπτύξουν το δυναμικό τους, να αυτό εκπληρωθούν και να έχουν μια ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία των πόλων με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές Πολλά μπορούν να προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εμείς στο EuroCities, στο δίκτυο ευρωπαϊκών πόλων, πιστεύουμε ότι πολλά έχουμε να κερδίσουμε από μια πιο συστηματική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών δήμων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μπιάνκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα δείχνει ότι στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας της έχει ένα από τα μεγάλα θέματα από το οποίο εξαρτάται το μέλλον της Υπήρου μας. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε, να εκφράζουμε γνωμοδοτήσεις και απόψεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα θέματα. Εδώ και κάποιες εβδομάδες στη Βόρεια Ιταλία ένα λεωφορείο που είχε προορισμό να πάει στο σχολείο παιδιά μιας μικρής πόλης ε, απήχθη από τον οδηγό του αυτοκινήτου το είδατε στις εφημερίδες φαντάζομαι που ήταν ένας μετανάστης στη χώρα μου βέβαια αυτή η εικόνα του εγχρώμου αυτού ανθρώπου που πήγαγε το Πούλμαν επικράτησε στις φωτογραφίες και δημιούργησε νέους φόβους μετά απεκαλύφθη ότι αυτό που μπορούσε να είναι μια τραγωδία, διότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε να βάλει φωτιά στο λεωφορείο, ήταν ένα από τα παιδιά που ήταν ε, στο λεωφορείο που ήταν, ε, γεννήθηκε στην Ιταλία και ήταν από γονείς ε, Αιγυπτίους. Ξεκίνησε μετά μια ευχαριστία Ευχαριστίε προ αυτό το παιδί που μετά ήθελε να γίνει αστυνομικό στα μεγαλώσει. Μιλάει τέλεια τα Ιταλικά, αισθάνεται Ιταλό και επέδειξε ότι είχε μεγάλο θάρρο που αντιμετώπισε το πρόβλημα και βοήθησε να σωθούν τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να διχαζόμαστε, Πρόεδρε, όσον αφορά τι πολιτικέ για την ένταξη. Αλλά στι πολιτικέ για τους μετανάστες είναι κατανοητό ότι έχουμε διαφορά. Στην Κατάνια, στην πόλη μου, έχουμε έναν καταλημμένο τόπο ε, τελικά τον ε, κάναμε ε, χώρο με κοινοτικά 20 παιδιά από τη Σικελία και 20 παιδιά από του μετανάστε εκεί καθάρισαν αυτό το χώρο, το μεταμόρφωσαν και είχαν συμφωνήσει και οι κάτοικοι. Διότι είδαν αυτά τα παιδιά να εργάζονται για ένα πρόγραμμα και είδαν ότι είναι θετικό αυτό. Καθάρισαν λοιπόν αυτό το χώρο. Αυτές είναι καλές πρακτικές που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. συνάδελφος Hans Janssen έχει το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Βαν Λάουερ θέλω να συνεχίσω κι εγώ. Υπάρχουν παραδείγματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εμείς έχουμε 8 συμβούλια που συνεργάζονται στην περιοχή μου. Συνεργαζόμαστε με άλλους που έρχονται στο κέντρο ασύλου και αναλαμβάνουμε τα άτομα που έρχονται, βλέπουμε ποιε είναι οι δεξιότητε που έχουν, διαρευνούμε τι δυνατότητε που έχουν να βρουν δουλειά στην περιοχή μα, καθώ και το ενδεχόμενο να βρουν στέγαση. Δηλαδή, ε, ε, προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις διάφορες ανάγκες. Είναι κάτι πιο χρονοβόρο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, όμως αυτό μέσω της προσωπικής αντιμετώπισης μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μακριά, εις βάθος χρόνου, μετά, όσον αφορά στο γραφείο μου, όταν καταφθάνουν άνθρωποι που έχουν ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή και δέχονται την Ολλανδική υπηκότητα, διότι έχουν βρει ότι υπάρχει διασύνδεση με τη χώρα, σύνδεσμος με τη χώρα, τότε αυτό είναι μια ικανοποίηση. Ε, και λένε αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε αυτή την κοινωνία. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία. Αν ε, δημιουργήσουμε πλατφόρμα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να μάθουμε τα διάφορα παραδείγματα που υπάρχουν και να μην βασιζόμαστε στην αρνητική άποψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη. Ε, συνάδελφε Ντεκώστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, λοιπόν, είμαι μέλο τη Επιτροπή των Περιφερειών επί Μακρόν και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που συνεχώ εξελίσσεται τα τελευταία 7 χρόνια. Ε, καταρχάς, οι περισσότερες τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή των Περιφερειών το ζουν το θέμα αυτό. Ε, δεν, είναι, δεν υπάρχει κάποια περιοχή που δεν έχει διερωτηθεί για το θέμα και δεν έχει διαβεί κάποιες αποφάσεις. Είμαστε στην πρώτη γραμμή πραγματικά σε αυτό το θέμα αυτό και βλέπουμε ότι είναι μια νέα μέθοδος που θα πρέπει να εφεύρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια νέα μέθοδο διότι αυτό το θέμα εξελίσσεται συνεχώς μεταλλάσσεται, η μετανάστευση αλλάζει γεωγραφικά, αλλάζει πλευρά ένταση και αλλάζει και προορισμού. Για απόδειξη βλέπουμε πώς άλλαξαν τα πράγματα στην κοινότητά μου του Σαντομέ, στην περιοχή μου. Ε, βρίσκομαι περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καλέ, όπου η κατάσταση άλλαξε ε, τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν διότι θέλουμε προφανώς να μπορέσουμε να προσφέρουμε δρόμους ένταξης στους μετανάστες, να φροντίσουμε ώστε οι κοινότητές μας να μπορούν να εξασφαλίσουν μια συνοχή μεταξύ των πολιτών αυτών που ζουν σε αυτή την περιοχή. Να, ήθελα να εκφράσω αυτή την εμπειρία της κοινότητάς μου που κάπως μαζέψαμε τους νέους γύρω από τον αθλητισμό. Στην κοινότητά μου νέοι Αυγάνοι, νέοι Πακιστανοί, συνοδευόμενοι από τους κατοίκους της ε, περιοχής και της πόλης μου θέλουν να δημιουργήσουν μια λέσχη κρίκετ. Ειδού λοιπόν όπου ο τελικό τη περιοχή εδώ και μερικέ εβδομάδε έφερε το Σαν Τομέρ 1 κατά Σαν Τομέρ 2 στο κρίκετ ε, ε, και όλες οι άλλες ομάδες μείνανε πολύ πίσω πρώτη δεύτερη θέση. Αυτές οι ομάδες που δημιουργήθηκαν λοιπόν ε, από νέους μετανάστες και επέλεξαν να δημιουργήσουν μια ακαδημία του κρίκετ για να ανοιχθούν αυτά, αυτές οι σχολείς προς τους άλλους ε, νέους και να μπορούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του κρίκετ να μοιραστούν κάποιε στιγμές. Λοιπόν, οι δύο μετανάστε που έγιναν πρωταθλητές και μετανάστες που γίνονται παράγοντες συνοχή και έτσι εδώ και ήθελα να ανταλλάξω μαζί σα μια καλή πρακτική. Ευχαριστώ πολύ. σου Σουμπίρα. Ευχαριστώ πολύ. Οι μεταναστευτικέ ροέ ε, αποτελούν μια πρόκληση που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Έχει και μια σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμω, οι αποφάσεις αυτές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν λαμβάνονται ή αναβάλλονται ή δεν έχουν, έχουν ε, την αναγκαία ευελιξία για να προσαρμόζονται στην κατάσταση η οποία αλλάζει συνεχώ. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας μεταξύ κρατών μελών να καταρρίξουν σε συμφωνία. Θέλω να εκφράσω λοιπόν την πεποίθησή μου ότι οι αρχές σε υποκρατικό επίπεδο είναι στρατηγική σύμμαχοι των ευρωπαϊκών θεσμών και των άλλων κρατικών αρχών που θέλουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την μεταναστευτική πρόκληση. Να σας δώσω παραδείγματα. Από τη μία έχουμε την πρόσταση ΣΕΡ που υπέβαλε η κυβέρνηση της χώρας των Βάσκων μαζί με άλλες περιφερειακές κυβερνήσεις που ε, βασίζεται στην ευθύνη της ε, ε, υπευθυνότητας. Share. κατανομή στα αγγλικά, ούτως ώστε να υπάρξει αναγκαία κατανομή ευθυνών. Η φόρμουλα αυτή είναι η διανομή λοιπόν των ευθυνών με βάση τους ε, πόρους, δεύτερον ε, τον πληθυσμό και τρίτον το ποσοστό ανεργίας. Με αυτή την πρόταση οι διάφορες υποεθνικές αρχές στέλνουμε και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την διάθεσή μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεύτερον, θέλουμε την ε, κοινοτική αιγίδα και κάλυψη. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για, μαζί με το ΑΚΝΟΥΡ και την Ισπανική κυβέρνηση. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την υποδοχή των μεταναστών και των οικογενειών του με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων και των συμπολιτών μα. Δεσμευόμεθα όλοι να προσφέρουμε για ένα ολόκληρο χρόνο οικονομική, κοινωνική και συναισθηματική στήριξη για να υποδεχθούμε και να βοηθήσουμε την ένταξη πέντε οικογενειών από την Υπεριορδανία. Ε, Έτσι βοηθάμε και την πρωτοβουλία πόλης και περιφέρειες. Να λοιπόν δύο παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι είμαστε τμήμα της λύσης. Άρα θα πρέπει να είμαστε τμήμα και της λήψης αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, επειδή έχουν ζητήσει πολύ το λόγο, 11 ακόμη, και γιατί πρέπει να σεβαστούμε το πρόγραμμα εργασιών μας, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουμε στις 6.30. Ο χρόνος ομιλίας είναι ε, από εδώ και στο εξή ένα λεπτό. Κίντο Βόλφο επομένως. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Δείχνει τι ε, πολύτιμος είναι ο ρόλος των ε, κοινοτήτων και των περιφερειών. Είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη και η προϋπόθεση είναι επίσης οι κοινέ μας αξίες που είναι ε, ο συνδετικός ιστός των κοινωνιών μας ούτως ώστε αυτοί που έρχονται αναμένουμε να σέβονται αυτούς τους κανόνες. Πρέπει λοιπόν να τους μάθουν. Στη Βάδη Βιρτεμβέργη Έχουμε αγωγή του πολίτου για τους ε, ετούντες άσυλο και μετανάστες όπου εργάζονται 300 δικαστές και δικηγόροι. Τους ενημερώνουμε για το κράτος δικαίου, τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους, για τις αξίες που αναμένουμε να τηρούν. Αυτό δείχνει τι δυνατότητες κρύβονται στην κοινότητά μας για μια επιτυχή ένταξη. Ελπίζω και σήμερα στην Επιτροπή Περιφερειών να συζητήσουμε για τέτοια επιτυχημένα προγράμματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιωάννα Μίκελ Λάιτνερ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι η ένταξη αρχίζει ήδη από τον υπηαγωγείο εδώ και μερικά χρόνια έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα όπου έχουμε και στα σχολεία ε, διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι γνωρίζουν 70 γλώσσες οι οποίοι φτιάχνουν γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των γονέων μεταξύ των παιδιών και των άλλων παιδιών αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει στη ζωή πόσο βοηθάει την ένταξη έτσι 20% των παιδιών μας στα νηπιαγωγεία που είναι μεταναστευτικής προέλευσης μπορούν να ενταχθούν και να βοηθηθούν από την νηπιαγωγείο μέσω αυτών των ε, διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και συνεργατών. Στην κάτω ε, Αυστρία έχουμε επιτύχει αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορεί να σας βοηθήσει και εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Από πλευρά μου δεν θα αναφέρω άλλα παραδείγματα παρά το ότι η πόλη μου, το Μάνχαεμ, 120.000 κατοίκων, εκ των οποίων 40% είναι μεταναστευτική προέλευση, θα μπορούσε πολλά παραδείγματα να αναφέρει. Αλλά να αναφέρω ορισμένα θέματα για, τις, ε, για τους Δήμους. Η πολιτική ένταξη και η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορούν να διαχωριστούν. Τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίζουν ούτως ώστε ένα τμήμα των ε, μεταναστών που δεν είναι σε θέση να ενταχθούν ε, στην αγορά εργασία γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση οι οποίοι κάνουν ζημιά στις κοινότητες μας. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο είναι υπάρχει αυτή η αντίληψη της ε, πόλης, των πόλεων άφηξης. Αλλά στην ουσία είναι γειτονιές άφηξη. Πρέπει να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη πολιτική για αυτές τις γειτονίες. Όχι μόνο για μετανάστες, αλλά για όλους του κατοίκου αυτών των ε, ε, περιοχών. Ευχαριστώ πολύ. Η Άννα Μαγκιάρ. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε πολύ που ο Επίτροπος ε, δέχτηκε με την πρόσκληση στη συζήτηση, αλλά με το που ξεκίνησε η συζήτηση έφυγε. Είχαμε μεταναστευτική κρίση χρόνια ολόκληρα στην Ευρώπη. Σε όλα μας τα εξωτερικά σύνορα. Παρόλο που πολλοί πολιτικοί ε, προτίμησαν να εθελοτυφλούν μπροστά στο φαινόμενο αυτό και να το αποσιωπούν. Και έχουμε ε, Πραγματικού πρόσφυγε, αλλά έχουμε και παράτυπου μετανάστες, εκατομμύρια, που είναι θύματα των εμπόρων, των λαθροδιακινητών, εμπόρων ανθρώπινων όντων και λαθροδιακινητών. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα και την τρομοκρατία. Η παράνομη μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το στήριξε όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, δίνονται τραπεζικές κάρτες στους μετανάστες μερικές φορές ε, τέτοιες ε, κάρτες χρηματοδοτούν την τρομοκρατία mm. τι έκανε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιστρέψουν οι μετανάστες στην πατρίδα τους και να βοηθήσουμε καλύτερα τις χώρες Ασίας και της Αφρικής να λύσουν τα προβλήματά τους αντί να εισάγουμε τα δικά τους προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχαριστώ Κυρία Μπεκόνια Μαρτίνες έχει το λόγο Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι με στην πολυμορφία και την πολυφωνία που παρατηρούμε έχουμε μια κοινή πρόκληση, την πρόκληση της μετανάστευσης. Και πολλές ε, περιφέρειες και δήμοι γνωρίζουν ότι είναι μεγάλη πρόκληση τη μετανάστευση. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο τη μετανάστευση και να περιλάβουμε σε αυτό τη διαχείριση τη πολυπολιτισμικότητα. Γιατί μιλούμε για πολυμορφία, για διαφορετικότητα, για πολιτισμικό πλούτο και το ανέφερε και ο επίτροπο προηγουμένω. Ακούμε όμω και πολύ ρητορική μίσου, πολύ μυσαλλοδοξία και έχουμε και άνοδο του λαϊκισμού. Γι' αυτό θα πρέπει και το δικό μα αφήγημα να είναι πιο θετικό, πιο συγκεκριμένο και χρειαζόμαστε άμεσε ενισχύσει όπω ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τοπικά προγράμματα και σχέδια και σε περιφερειακέ πρωτοβουλίε που προωθούν αυτά τα νέα μοντέλα διακοινωτικής επικοινωνία και δημιουργούν διάβλους διαλόγου, συμμετοχής και χειραφέτηση του πολίτη και ιδιαίτερα των μεταναστών. Αυτά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αλφόνσο Πλεγουεσουέλο. Ευχαριστώ. Μιλούμε για ένταξη. Η ένταξη είναι ακρογωνίως λήθος της πολιτικής για την Ευρώπη το 2020. Θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, ανήκει ε, και στην ατζέντα του 2030 και στους βιώσιμους, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα πίσω. Κατάγομαι από τη Μούρσια, που είναι από τις παράκτητες περιοχές ε, της Ισπανίας, ε, στην Νότια Μεσόγειο και έχουμε συνηθίσει να υποδεχόμαστε μετανάστες πολλές φορές είναι και παράτυποι αυτοί οι μετανάστες. Αυτό που μας προβληματίζει όμως και που μας απασχολεί είναι ότι ε, όσο συντονίζουμε την πολιτική υποδοχής και τη πολιτική της μετανάστευσης να συντονίζουμε και τις πολιτικές γιατί γίνεται μετά την άφηξη γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο η υποδοχή, η φιλοξενία αλλά και η ένταξη. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας βράβευσε με ένα ευρωπαϊκό βραβείο χάρη στα προγράμματα επαγγελματικής ένταξης των μεταναστών γιατί πιστεύω ότι η απασχόληση είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική γιατί χωρίς ε, επαγγελματική ένταξη δεν θα επιτύχουμε την κοινωνική ένταξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλαμπουίκ. Θα μιλήσω στα καταλανικά. Αυτό μιλάμε στην Βαλένθια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ καταρχήν που διοργανώσατε αυτή τη σημαντική συζήτηση και τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Πρόκειται για ένα κέριο ζήτημα. Και όπως είπαμε, οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την υποδοχή, φιλοξενία και ένταξη των μεταναστών. Και γι' αυτό θα ήθελα να προσυπογράψω και εγώ όλα αυτά που είπαμε και τα αιτήματά μας. Το είπε και ο Επίτροπος. Αν αυξηθούν τα κονδύλια, σίγουρα και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να γίνουν οι αποδέκτες αυτών των αυξημένων κονδύλιων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε όλο και περισσότερους ασυνόδευτους ανηλίκους ε, μετανάστες, όλο και περισσότερους. Και αυτοί οι ανήλικοι είναι πια μια πολύ σημαντική ομάδα. Μιλούμε για χιλιάδες ασυνόδευτους ανηλίκους. Θα πρέπει ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες, να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία και την μυσαλλοδοξία ή το μίσος κατά των φτωχών. Και αυτό που είπε η κυρία προηγουμένω, που συνέντεσε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία, το θεωρώ άθλιο και ελεηνό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο αποκλεισμό δημιουργεί πρόσφορο έδαφο για τη ριζοσπαστικοποίηση. Οπότε μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση χάρη σε μια πολιτική ανάπτυξη που θα περικλεί, που δεν θα αποκλεί κανένα ανάπτυξη για όλου, όπω λένε και όσα. Και πολλές άλλες οργανώσεις. Είχαμε 40.000 ε, ε, μετανάστες από 38 χώρες, 10% της ε, δικής μου πόλης. Έχουμε ένα σχέδιο υποδοχής και ένταξης, αλλά περισσότερο από ένταξη αυτό που θέλουμε είναι συμβίωση, συνύπαρξη με σεβασμό της διαφορετικότητας, της πολυμορφίας και με την πλήρη ένταξη των μεταναστών. Η μετανάστευση είναι πλούτος ε, για την αγορά εργασίας, για τη δημογραφία, για τις διαπολιτισμικές ε, ε, συναλλαγές και επαφές. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η ένταξη συνάδει με το μοντέλο μας, το κοινωνικό μοντέλο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης για όλους. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Πολίνα Χαϊάννεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην περιοχή μου στην νοτιοτιδική Φιλανδία έχουμε διοργανώσει μαθήματα για οικογένειες μεταναστών για τις μητέρες των οικογένειών διότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους οι μητέρες μαζί τους να κάνουν μαθήματα φιλανδικών μπορούν να κάνουν μαθήματα που αφορούν την κοινωνία της Φιλανδίας, να μάθουν τους κανόνες που ισχύουν, πώς μπορεί να υπάρξει μέρημνα για τα παιδιά κλπ. Διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Ε, όλα αυτά εφαρμόζονται λοιπόν αυτά στην περιοχή μας. Έχουμε τελικά τύχη μεγάλης υποστήριξης και βοηθήσαμε τελικά στις γυναίκες να μπορούν να φύγουν από τους τοίχους του σπιτιού και να μπορούν να συμμετάσχουν στην ενεργό ζωή της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Πελ Γκραντφαλτ, ο συνάδελφος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάνω σε αυτά που έθιξαν συνάδελφοι θέλω να πω και εγώ κάτι. Μίλησα για την ανάπτυξη. Εγώ είμαι υπεύθυνο μια τοπική αρχή που έχει 30% των κατοίκων που έχουν γεννηθεί στην Αλοδαπή. Είναι πολλούς μετανάστες η περιοχή μου σε σχέση με άλλες τοπικές αρχές. Έχουμε μόνο 8,5% επίπεδο ανεργίας. Και όπως είπαν πολλοί, το κλειδί είναι ότι δημιουργούνται ε, τοπικά θέσει εργασίε με υψηλού ρυθμού ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπω είπε και ο Επίτροπο, υπάρχουν πολλά τέτοια καλά παραδείγματα. Πρέπει να τα αναφέρομαι. Χαίρομαι που διεξάγεται σήμερα αυτή η συζήτηση, διότι η ανάπτυξη είναι ένα από τα κλειδιά για να εξασφαλίσουμε την ένταξη. Να μπορεί να λειτουργήσει η ένταξη. Χαμηλή ανεργία, κυρίως για εκείνους που γεννιούνται στο εξωτερικό και για τους μετανάστες, βοηθά την ένταξη. Και είναι πολύ καλό που διεξάγει τη συζήτηση και μπορούμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ντονάτο Τωμά, ο συνάδελφος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ντονάτο Τόμε. Ε, είμαι νομάς περιοχής του Μολίζε θα ήθελα να αναφερθώ στη θετική εμπειρία της περιοχής του Μολύζε. χιλιάδες μετανάστες περίπου ε, δέχτηκαν, 300.000 οι κάτοικοι. Είναι σωστός αριθμός, αυτό που σημαίνει ότι κάποια τα μυστικά για να γίνει σωστή υποδοχή, αξιοπρεπής υποδοχή, αξιοπρεπής λέγω προσοχή, είναι θεμελιώδης λέξη αυτή για την υποδοχή, διαφορετικά σημαίνει κάτι άλλο και συσχετισμό αριθμού μεταναστών με τον πληθυσμό υποδοχής και κατανομή των μεταναστών στην περιοχή είναι κάτι σημαντικό. Για την ένταξη να προσθέσω αυτό που ήδη υπόθηκε ότι το Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζει πολλά προγράμματα, πολλά προγράμματα στο σχολείο για την ένταξη των αμφιχθέντων και επίση και οι ενορίε κάνουν πολλή δουλειά σε εμά, διότι είναι παρούσε οι ενορίε και στην υποδοχή και στην ένταξη των μεταναστών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίος. Μιλάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έλλειψη της ένταξης δημιουργεί περιθεριοποίηση και παράγει φτώχεια από την περιθυροποίηση μέχρι τη φτώχεια, από αυτά γεννιέται, γεννιέται και ο ρατσισμός. Αλλά χρειάζεται μια πανέμβαση εκεί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να πανέμβουμε. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να παίξουν ρόλο οι τοπικέ αρχέ. Θετικά χαιρετίζουμε αυτά που είπε ο Επίτροπο. Θα υπάρξουν πόροι, είπε. Δεν αρκούν όμω. Και δεν αρκούν, ξέρετε γιατί. Διότι θα πρέπει έναντι μια πολύ μεγάλη μετανάστευση ε, πρωτοφάνου που αποτελείται και από νόμιμους μετανάστες και από λαθρομετανάστες. Όμως οι λαθρομετανάστες είναι αυτοί που δεν καταφέρνουν να μπαίνουν με το σωστό τρόπο, με τον νόμιμο τρόπο στην επικράτειά μας. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν τους σταματήσουμε απλώς βοηθώντας τους ε, ε, στην πατρίδα τους εκτός Εάν η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει πραγματικά να αλλάξει τα χαρτιά της τράπουλας και να δώσει πόρους, πολλούς πόρους για να βοηθήσει στην πατρίδα τους αυτούς. Μόνο με πολλούς πόρους μπορούμε να βοηθήσουμε στις πατρίδες τους. Διαφορετικά είναι ένα σύνθημα διαφημιστικό που θα μας ε, ε, θα οδηγήσει στο να μας κατακλείσουν τελικά εκατομμύρια ανθρωπινά που θα καταφτάσουν επικράτειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, τους και τις συναδέλφους. Και πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Μαντζινέλη για να κλείσει τη συζήτηση από πλευρά τη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από όλε τις παρεμβάσεις θεωρώ ότι διαφαίνεται ένα πανόραμα, μια γενική εικόνα που μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. Εμείς σαν πόλη, σαν πόλη της Αγκώνας σε δύο χρόνια, για δύο χρόνια οργανώνουμε ένα φεστιβάλ κάθε χρόνο. Σε μια από τις συνοικίες της πιο πολυεθνικές της πόλης, όπου οι πολίτες ε, της Αλοδαπής είναι 30 με 40% του πληθυσμού που διαμένει εκεί, είναι ένα φεστιβάλ που θέλουμε να γίνεται μια ευκαιρία κάθε χρόνο για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και όλο και περισσότερο να γίνεται έτσι. Να είναι ένα είδος εργαστήριο ε, για να μπορεί να γίνεται ανταλλαγή μεταξύ εκπροσώπων τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένων καλών πρακτικών. Όχι αυτά που αναφέρονται στο συνέδριο. Πραγματικέ πρακτικέ που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δράτε με τι ευκαιρίε να καλέσω όλου σα σε αυτή την πρωτοβουλία που όποιο ενδιαφέρεται και να διασυνδεθούμε για να ανταλλάξουμε απόψεις και εκτός ε, του, της Επιτροπής των Περιφερειών με τις πρακτικές. Και να αναφέρω κάποια τελική σκέψη πάμε σε όλα αυτά. Από όλε τι παρεμβάσει και από τι εμπειρίε που έχουμε ο καθένα από εμά, βλέπουμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε ένα μάθημα. η αριθμοί είναι κάτι σημαντικό. Οι αριθμοί, η ποσότητα και οι άνθρωποι που καταφθάνουν και η, ποιότητα των, η ποσότητα των διαθέσιμων πόρων, οι καλές πρακτικές. Τα εκατομμύρια στον κόσμο μπορούν να λειτουργήσουν σε κάποια επίπεδα και να μην λειτουργήσουν αν οι αριθμοί ε, των αποδεκτών των βέλτιστων πρακτικών και οι αριθμοί των διαθεσίμων πόρων, τα ποσά αυτά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Αν φτάσουν σε μια πόλη 100.000 κατοίκων σε ένα χρόνο περιορισμένο 1500 άτομα που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι τα πάντα. Σπίτι, δουλειά, να μιλήσουν τη γλώσσα. 1500 άτομα δεν μπορεί να τα εντάξεις με λίγα χρήματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν φτάσουν 3000 δεν μπορείς κανέναν να εντάξεις. Λοιπόν, οι καλές πρακτικές και οι αρχές είναι θεμελιώδεις, αλλά αν μετά δεν κάνουμε λογαριασμούς και δεν λάβουμε υπόψη τα νούμερα, πιστεύω ότι και οι καλές πρακτικές και οι καλές αρχές κινδυνεύουν να παραμείνουν μόνο επί χάρτου. Καλή δουλειά σε όλους σας και ελπίζω να σας συναντήσω σε μια επόμενη ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαντσινέλη. Ευχαριστώ για την ε, καλή σας πρακτική. Το παράδειγμα που δίνετε στην πόλη σας. Ελπίζω να εμπνεύσει και τη δική μας πρωτοβουλία για την ένταξη των μεταναστών. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και άλλες πόλεις αλλά 83 που ήδη έχουμε δεν είναι και λίγε. Καλή τύχη. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα περνάμε στο 5 της σημερινής διάταξης. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την Πολιτική Συνοχής και η προσαρμογή των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Παρακαλώ τον εισηγητή μας κύριο Ρόμπ Γιόγκμαν να έρθει εδώ στο Προεδρείο μαζί με τον εμπειρογνώμονά του και χαίρομαι που μπορώ να σας ε, ανακοινώσω ότι και η κυρία Μιχαήλοβα, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμμετάσχει στη συζήτηση you and thank you for the Thank you Sans tarder, je donne la parole. Λοιπόν, το λόγο εισηγητή Thank you very much, uh, Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μιχαήλοβα για την παρουσία της. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Δεν θέλω να σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά το θέμα είναι τεχνικό. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότησης που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας. Είναι αρκετά καλό το Ταμείο Συνοχής ή τα Ταμεία Συνοχής είναι αρκετά ευέλικτα και πώς μπορούν να συμμετάσχουν καλύτερα οι περιφέρειες ε, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Να λοιπόν ποιες είναι οι βασικές αρχές. Επικουρικότητα, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και συνεργασία. Η πολιτική συνοχής ε, βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα τρία στοιχεία. Και υπάρχει και ένας κώδικας διοντολογίας που το καθορίζει αυτό. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εγγυάται αυτά τα τρία στοιχεία. Εγγυάται ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Και είχα εκπονήσει κάποτε και μία γνωμοδότηση για, το ευρωπαϊκό, για τον κώδικα δοντολογίας και για τη σύνδεση των περιφερειών και κοινοτήτων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά δεν την ενθουσίασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα η γνωμοδότησή μας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το χαιρέτησε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η πολιτική συνοχή και το ευρωπαϊκό εξάμεινο να συνδυάζονται καλύτερα. Γι' αυτό οι κοινότητε και οι περιφέρειε πρέπει να συμπεριληφθούν ακόμη περισσότερο τώρα πλέον. Το 2017 εκφράσαμε αυτή την επιθυμία μας στον κώδικα διοντολογίας και εξακολουθεί να ισχύει το αίτημά μας. Τώρα λοιπόν θέλουμε να συνδυάσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο δηλαδή τα επόμενα ευρωπαϊκά εξάμεινα για την περίοδο 21-27 με το πολιτές πλαίσιο. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο η συνεργασία και ο κώδικας δοντολογίας όλα αυτά συνδυάζονται. Βασική αρχή είναι ο κώδικα διοντολογία να εφαρμόζεται πολύ περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε αυτό μα στηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στι εκθέσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά χώρα για το 2019 υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει για την ε, εκταμείευση των πόρων συνοχή για την περίοδο 21-27. Θα το δείτε στο παράρτημα. χρειαζόμαστε κάποια εγγύηση ότι οι κοινότητες και οι περιφέρειες θα συμμετάσχουν. Οπότε ενέκρινε το αίτημά μας και η ε, Ρουμανική Προεδρία. Εάν οι περιφέρειες και οι κοινότητες θέλουν να συμμετάσχουν ήδη από την προπαρασκευαστική φάση στην εκπόνηση της ε, πολιτικής συνοχής αυτό πρέπει να επιτραπεί. Και νομίζω ότι το εγγυάται ο νέος κανονισμός. Υπευλήθησαν κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ τι πολιτικές ομάδες Του σοσιαλιστές και άλλους που συνεργάστηκαν δεν μπορώ να τη στηρίξω όμω όλες τις τροπολογίες γιατί γιατί μόνο το σενάριο 1 επιτρέπει την ε, συμμετοχή των περιφερειών και κοινοτήτων. Ε, συμπαθητικό αυτό. Αλλά νομίζω ότι οι επόμενοι συντάκτες ε, εκθέσεων θα έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε τις αποφάσεις που θα λάβουν εκείνη τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, χαίρομαι ε, για την ε, ότι υπάρχει ε, συμφωνία μεταξύ μας, έτσι ενισχύεται το μήνυμα που στέλνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω αυτόν που κάθεται δίπλα μου, την κυρία που κάθεται δίπλα μου, που συνεργαστήκαν πολύ στενά. Ευχαριστώ την πρόεδρο, την κυρία Μιχαήλοβα, η οποία παρουσίασε μια γνωμοδότηση την οποία υποστηρίζω πλήρως και ελπίζω η υποστήριξη να είναι αμοιβαία. θα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Κοτέρ, τους ε, εκείνους που εργάστηκαν στην Επιτροπή, τους ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία, ευχαριστώ επίσης τη γραμματεία της Επιτροπής ΕΚΟΝ, τον κύριο Φορ, α κάπου εκεί, ευχαριστώ Ανδρέα είσαι εκεί στη γωνία, έκανες πολύ καλή δουλειά και μετά τη γραμματεία της ομάδας μου, το Γιάκομπ, ευχαριστώ Γιάκομπ, ε, φαίνεται σαν να είμαστε στα Όσκαρ, στην τελετή των Όσκαρ με όλε αυτέ τι ευχαριστίε. Όμω αξίζουν τι ευχαριστίε, γιατί πραγματικά είχαμε πλήρη υποστήριξη από του συνεργάτε και από πλευρά πολλών τοπικών φορέων. Και μετά θέλω να ευχαριστήσω και τον εμπειρογνώμονά μου, τον κ. Βαν Μπόρχ, που κοκκινίζει τώρα αλλά του αξίζει ε, η ευχαριστή αυτή. Τον ευχαριστώ για την υποστήριξη και την πρόσκληση στο γεύμα χτες ε, το βράδυ. Όχι, όχι. Εντάξει, αστείευομαι τώρα. Ε, χαίρομαι που συνεργαστήκαμε μαζί. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη συνεργασία. Ευχαριστώ. Λαμπρά. αλλά Τις ευχαριστήσω να τι κάνετε εντό του χρόνου αγόρευσή σας. Ε, εσείς τις κάνετε εκτός και ξεπεράσετε το χρόνο κατά 1,5 λεπτό και θα ακούσουμε τώρα την πρόεδρο τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ίσκρα Μιχάηλοβα. Και θα ήθελα επ' να την ευχαριστήσω θερμότατα για την ε, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια τη κοινοβουλευτική θητεία μαζί της και με την Επιτροπή, που, με την Επιτροπή Ρέγγι, την Επιτροπή Περιφερειακής Και είδαμε και ε, πολύ απτά αποτελέσματα αυτής της αγαστής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ κυρία Μιχαήλοβα και σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση να συμμετάσχω σήμερα εδώ και να σας παρουσιάσω την ε, άποψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, για την ε, συζήτηση που γίνεται για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Τον περασμένο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμά του για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη για το 2019 που επιβεβαιώνει και πάλι την ε, ανάγκη αύξησης ποιοτικών επενδύσεων, ε, μεταρρυθμίσεων και στήριξη της ε, αύξησης της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης για όλους και της μακροχρηματοοικονομικής σταθερότητας και της εξηγήσης των δημόσιων οικονομικών. Επίσης, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να λάβουν αποφασισμένες και συντονισμένες δράσεις, ώστε να υλοποιήσουμε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Επίσης, ε, δίνουμε έμφαση στην ανάγκη αύξηση παραγωγικότητας από τα κράτη-μέλη με αύξηση των επενδύσεων. Επενδύσεις πρέπει να δίνονται στην ανάπτυξη και σε σχέδια βιώσιμων υποδομών με βάση τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και του ΟΗΕ και ε, προσπάθεια τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Αύξηση τη παραγωγικότητα, προποθέτει επίση επενδύσει στι δεξιότητε, στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, στη βιώσιμη κινητικότητα και τι αντίστοιχε υποδομέ με βάση του στόχου τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που μπορεί να γίνει με κονδύλια τη πολιτική συνοχή ε, σε συνέργεια όμως και συμπληρωματικότητα με άλλα κοινοτικά προγράμματα και μηχανισμού. Η αύξηση της παραγωγικότητας και η απάταξη των αποκλεισμών θα πρέπει να είναι κοινό στόχος των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών αλλά και των μεταρρυθμίσεων των περιφερειών. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη γνωμοδότησή της ε, που είχα την τιμή μάλιστα να συντάξω εγώ τονίζει ότι η καλύτερη εστίαση σε επενδύσεις της πολιτικής συνοχής και στη συμπληρωματικότητα με τα άλλα κοινοτικά προγράμματα είναι απολύτως απαραίτητα. Επίσης, χρειαζόμαστε και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους και να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να προσελκύσουν και δημόσιες αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις, να προωθήσουν συμπράξεις σε δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ζητούμενο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των κονδυλίων ε, της ε, συνοχής και της συμπληρωματικότητα του με τι άλλε πολιτικέ τη Ένωση. Από αυτήν την άποψη τα μέλη τη Επιτροπή Ρέγκη καλωσορίζουν την πρόταση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και την ενίσχυση τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη ε, Πολιτική συνοχή, ώστε να επιτύχουμε ε, έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη για όλου. Επίση, ε, χαιρετίζουμε τη μεγαλύτερη έφαση που δίνεται από το οικονομικό εξάμεινο στι επενδυτικέ ανάγκε, με το νέο παράρτημα για τι επενδύσει στι εκθέσει αναχώρα και έτσι εντοπίζονται οι τοπικές και εθνικές ανάγκες επιδετικές σε σχέση με τα κονδύλια της συνοχής. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ελαστικότητα στην κατανομή των ευρωπαϊκών κονδύλιων, ώστε τα σχέδια των στρατηγικών επενδύσεων και τα σχετικά κονδύλια να πιάνουν τόπο. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ε, εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, με στόχο τη συνολική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ε, χάρη της ε, ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Εν ώψη των μελλοντικών διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων θα πρέπει να ενισχύσουμε την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως αναφέρει και ο εισηγητής σας αλλά και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που είναι απαραίτητη για τη βελτίωση όλων των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μέσω της επενδυτικής πολιτικής και μέσω της υλοποίησης πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα εξασφαλίσει ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή των ειδικών συστάσεων αναχώρα στην, και στην επενδυτική διαδικασία και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εν τέλει θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία μας με την Επιτροπή των Περιφερειών στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θετία ήταν εξαιρετικά καρποφόρα, επικοδομητική και έγινε σε πολύ θετικό κλίμα. Ακόμη και σήμερα είχαμε πολύ εθαρρυντική συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ τη πολιτική εδαφική συνοχή και προπολογισμού τη Ένωση. Και ελπίζουμε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και μετά τι ευρωεκλογέ με το νέο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ και πάλι για την αγαστή συνεργασία και για την ευκαιρία που μου δώσετε να σα παρουσιάσω τη γνωμοδότηση Επιτροπή Ρέτζι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινά λοιπόν η γενική μου συζήτηση. Έχω μόνο ένα αίτημα για παρέμβαση. Στο συνάδελφο φλεγό δίνω το λόγο, αν και άλλοι θέλουν να παρέμβουν, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν. Παρακαλώ. Ο κ. Φλεγού έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Μιχαήλοβα, κύρια Ισηγητά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε για αυτή τη συζήτηση και να ε, εγκομιάσω ιδιαίτερω την πολύ αξιόλογη γνωμοδότησή σα. πρέπει να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα σαφέ μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, αλλά και σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του σημερινού και του μελλοντικού. Και γιατί τα λέω αυτό, Γιατί εδώ εκπροσωπώ την Ίστρια, την πιο ανεπτυγμένη περιφέρεια της Κροατίας και πιστεύω ότι ε, έχει δείξει η Ιστρία πόσο προχωρεί και πόσο πιο ανεπτυγμένη είναι από την υπόλοιπη Κροατία. Μπορούμε να μιλούμε για κατακεφαλήνα ΕΠ, μπορούμε να μιλούμε για πολύ καλή δημογραφική εικόνα και για πολυάριθμα σχέδια και προγράμματα που έχουμε ετοιμάσει στην Ίστρια και θα υποβάλουμε για να λάβουμε κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα τονίσουμε και να τα εξάρουμε. Γιατί χάρη στην ανάπτυξη που διαπιστώνουμε καθημερινά στην Ίστρια και χάρη στις προσπάθειες και τη δομή της οικονομίας μας, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να συνδέσουμε τους μεγάλους επενδυτικούς μηχανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να τις συνδέσουμε ε, με τη με το Ζάγκρεπ, την πρωτεύουσα τη Κροατία. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τι επενδυτικέ επενδυτικές μεταξύ Βρυξελών και Ζάγκρεπ. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ του αποκεντρωμένου μοντέλου των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και η Ιστρία, όπω και οι υπόλοιπε περιφέρειε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να περιορίζονται από τι εθνικέ στρατηγικέ. Γιατί μερικέ φορέ οι εθνικές στρατηγικές ε, είναι άσχετε με τι τοπικέ του ανάγκε, και μερικέ φορέ αντιστρατεύονται τι τοπικέ ανάγκε οι εθνικέ στρατηγικέ ό,τι αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, η πολιτική συνοχή και η, σύνδεσμό τη με το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα περιορίσει το τοπικό δυναμικό. Αυτό θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Θα πρέπει αντίθετα να ενισχύσουμε τις περιφέρειες και τους Δήμους. Γι' αυτό και είμαι υπέρ της γνωμοδότησης και ε, συμμερίζομαι την έκκληση του εισηγητού να συμπεριληφθούν οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες στη δημιουργία των, των εθνικών πολιτικών από τη φάση της σύλληψης και χάραξης και στη φάση της εφαρμογής και με την αίσθηση κοινή ευθύνη σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης να εφαρμόσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γκαετάνο Αρμά, συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ σχετικά με ένα σημείο φορά την περιοχή μου, τη Σικελία, που ανήκει στι νότιε περιοχέ της Ιταλίας. Σε αυτό το τμήμα της χώρας, που είναι και το φτωχότερο τη Ιταλία, όπως αναφέρθηκε ήδη, από το Σφίμετς που είναι σημαντικό ίδρυμα ερευνών της Νότιας Ιταλίας και διάφορα λογιστικά της περιοχής. Το 2018 είδαμε ότι οι επενδύσεις οι δημόσιες οι κρατικές έχουν καταρρεύσει. Ενώ βλέπουμε αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Αυτή είναι η εικόνα. Άρα πρέπει να σημειώσουμε εδώ την αναγκαία ε, προσθετικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Σε κάποιε χώρε, μεταξύ αυτών και η Ιταλία και κυρίω περιοχέ τη Νότια Ιταλία, εφαρμόζουν ένα κριτήριο που αντικαθιστά αυτό του πόρου. Θα πρέπει να κάνει ελέγχου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να μην υπάρχει αντικατάσταση των ευρωπαϊκών πόρων με του κρατικού πόρου. Τα στοιχεία τη υπηρεσία μα τη λένε ότι οι δαπάνε για επενδύσει ήταν 28,9% του Ιταλικού κράτου στο Νότο, με μία μείωση ε, το τελευταίο τριετία 28,4%. Στη Βόρεια Ιταλία αυξάνονται οι επενδύσει σε συνάρτηση με τον πληθυσμό. Ο Ιταλός νομοθέτης έπρεπε δια νόμου να βάλει ένα όριο ελάχιστο. Όριο, ένα κατόφλιο κάτω από το οποίο δεν θα μπορούν να πάνε οι επενδύσεις στην νότια ε, Ιταλία σε σχέση με τον πληθυσμό διότι υπάρχει ασυμμετρία μεταξύ κρατικών επενδύσεων και πληθυσμού. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία τους επόμενους μήνες να εγγυηθούν το κριτήριο της προσθετικότητας όσον αφορά τις περιοχές της Νότιας Ιταλίας. Δεν είναι κάτι που απαιτούν οι κανονισμοί, αλλά είναι κάτι το, για το οποίο υπάρχει εγγύηση και απέτηση εφαρμογή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλος που να επιθυμεί να παρέμβει στα πλαίσια της γενικής συζητήσεως, οπότε φτάνουμε στην εξέταση των τροπολογιών. Τροπολογία 1 του εισηγητού που αντικαθιστά την τροπολογία 1 την αρχική. Ποιος είναι υπέρ? Α, ζητώ συγγνώμη. Αλμπέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σωστά ο εισηγητής λέγει ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα υποβάλει γνωμοδότηση σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού. Σχέδιο της νομοδοτήσεως όμως δεν συμπεριλαμβάνει την τροπολογία που προσπάθησε να συμπεριλάβει το κόμμα του Σελιστικού στο σημείο 7 της γνωμοδότησης του συγητού που έχει κατατεθεί μπροστά μας. Το να εγκρίνουμε αυτό το τμήμα της τροπολογίας του Σελιστικού Κόμματος που απέρριψε ο εισηγητής θα βοηθούσε να, λάβει, να ληφθεί υπόψη αυτό που θέλουμε να τονίσουμε. Βλέποντας αυτό που έχει απορριφθεί από τον εισηγητή στην τροπολογία του, εκεί μιλάμε για μακροπρόθεσμη μακροπρόθεσμο οικονομικό μοντέλο. Ο τίτλος νομοδοτήσεως είναι ευθυγράμμιση των θεωτικών μεταρρυθμίσεων με μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Με άλλα λόγια. Εκφράζουμε άποψη που είναι και ο τίτλος της νομοδοτήσεως που έχει κατατεθεί. Τελικό σχόλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο το ίδιο στις 26 Μαρτίου, δεν μιλώ για Επιτροπή, μιλώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο, που υιοθέτησε στη δήλωσή του ένα σημείο ή σειρά σημείων που αντικατοπτρίζουν την τροπολογία που προσπαθούμε να εγκρίνουμε εδώ τώρα. Για αυτούς τους προαναφερθέντες τρεις λόγους προτείνω να, απο, να απορρίψουμε τη θέση του εισηγητού και να θετήσουμε την τροπολογία ως κατετέθη από την ομάδα τη Σοσιαλιστική. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γενέντε Χέαρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αντίθεση με αυτά που λέει ο συνάδελφος Μπορ, Όσον αφορά την Ολλανδική αντιπροσωπεία, θεωρούμε σημαντικότατο ότι εάν ετοιμάζονται κάποιες εισηγήσεις στην Επιτροπή των Περιφερειών που μας δίνει δυνατότητα επιλογής, είναι σκόπιμο να περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα κείμενα. Γι' αυτό το λόγο τα μέλη της Ολλανδικής Αντιπροσωπείας θα υποστηρίξουν τον εισηγητή. Θέλει να απαντήσει μήπως ο κύριος ηγητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Φαντάζομαι, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Μπορ, αλλά είναι πολύ πρόημο τώρα να ληφθεί απόφαση. Um, δεν είναι ότι διαφωνώ με αυτά που μας είπε, αλλά δεν θα ήταν σοφόν, uh, ούτε κομψόν, uh, Ήδη τώρα να εγκριθεί τροπολογία 1. Δεν διαφωνούμε ουσιαστικά όσον αφορά το περιεχόμενο. Διαφωνούμε επί του χρονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Να ψηφίσουμε. Στην τροπολογία του εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Κατά. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Le Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία. Τροπολογία 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται πριν την τελική ψηφοφορία να διορθώσω ένα λάθο. Δεν έδωσα προηγουμένω το λόγο στην κυρία Πρόεδρο για να αντιδράσει στην ε, συζήτηση. Οπότε του δίνω συντόμω. της δίνω συντόμω το χρόνο και το χρόνο και της το συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα να αντιδράσω. Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις ε, τις οποίες βρίσκω σαν άξιες Νομίζω ότι το αίτημα της Ρουμανικής Προεδρίας να λάβει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών είναι πολύ σημαντική. Γιατί έτσι ακούγεται η φωνή της Επιτροπής Περιφερειών και το Συμβούλιο θα καταλαβαίνει πολύ καλύτερα πώς είναι η κατάσταση εν ώψη των ε, επικειμένων διαπραγματεύσεων για το μέλλον των επενδύσεων στην Ευρώπη και θα έχει και τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του συντάκτη της γνωμοδότησής σας και νομίζω ότι είναι και κατάλληλη στιγμή για να υποβληθεί η γνωμοδότηση αυτή. Όλοι πρέπει να είμαστε πιο δεκτικοί, πιο ευέλικτοι για να προσαρμοστούμε στις αλλαγές που καθημερινά επισυμβαίνουν για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τον νέο τρόπο επενδύσεων στην Ένωση αλλά να διατηρήσουμε και όσα θετικά υπήρξαν στο παρελθόν και η Επιτροπή Περιφυρών μπορεί ακριβώς να ε, είναι η φωνή της αληθείας. Έχουμε την, ε, τις θετικές εμπειρίες, τις καλές πρακτικές και όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων που όλοι επιθυμούμε. Σας συγχαίρω λοιπόν για την εργασία σας και ελπίζω και η Ολομέλεια να στηρίξει τη γνωμοδότηση αυτή στην τελική ψηφοφορία και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να λοιπόν που φτάνουμε ακριβώς στην τελική ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Να συγχαρούμε τον εισηγητή. Και να τον ευχαριστήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας με το επόμενο θέμα, τη συζήτηση για την πορεία προς έναν μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας. Βέβαια είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Τι θα πει ανταποκρίνεται και ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας, τι θα πει φιλοδοξίες. Και αυτό θα μπορούσε να μας απασχολήσει μια μισή ώρα αν συζητάμε αυτά τα θέματα, τι σημαίνει το ένα και τι το άλλο. Πάντως για αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ζαν Αχτουή, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση για να συζητήσουμε μαζί το μέλλον του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο θα δείξει ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας και συνοχής των κρατών μελών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να πούν χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα παιδιά μου θα ζουν το ίδιο καλά, ίσως και καλύτερα από μένα. Το ισχύον ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο ήταν χαμηλότερο από το προηγούμενο και σήμερα λόγω του Brexit φοβόμαστε ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Και τη στιγμή που έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη την Ευρώπη, δυστυχώς ε, τα κονδύλια δεν ακολουθούν τις προκλήσεις και ακόμη χειρότερο μπορεί να μειωθούν κιόλα. Και όταν όλες οι μελέτες δείχνουν ε, αύξηση των χασμάτων μεταξύ στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο τους Ευρωπαίους που χρειάζονται τέτοια κονδύλια όπου και αν βρίσκονται. Χωρίς οικονομική συνοχή, χωρίς εδαφική και κοινωνική συνοχή δεν θα έχουμε μια ουσιαστική ένωση. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να στηρίζει και την περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό το νόημα έχει η συμμαχία μας για τη συνοχή που έχει συγκεντρώσει σήμερα 12.000 ε, προσφορές, συνεισφορές που ε, είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των οργανώσεων. Και όταν μιλώ για υποστήριξη, εννοώ ότι το προπολογισμό αλλά και του δημοσιονομικού κανόνε που θα πρέπει να προσαρμοστούν για να απελευθερώσουν τι τοπικέ και περιφερειακές επενδύσει που χρειάζονται τόσο πολύ οι Ευρωπαίοι πολίτε. Κύριε Πρόεδρε, με τι ψηφοφορίε για το πολίτε, δημοσιονομικό πλαίσιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μα, ε, διαφαίνεται ένα κοινό όραμα των ερετών ε, της Ευρώπης και των ερετών των τοπικών και περιφερειακών αρχών για το μέλλον του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι μελλοντικέ επενδύσεις θα πρέπει να βρεθούν στο κέντρο το προβληματισμό μας, ιδιαίτερα με την πρόταση της Επιτροπής μας για, μια, για έναν ριζικό επαναπροσανατολισμό της κοινή γεωρικής πολιτικής, τη διαφύλαξη μιας ισχυρής και απλουστευμένης ε, πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων με εδαφικό προσανατολισμό και τον τριπλασιασμό του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα Έρασμος. Δυστυχώς όμως αυτή η σύγκληση που διαπιστώνουμε μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής των Περιφερειών δεν αντικατοπτρίζεται στο Συμβούλιο που ήδη έχει αναβάλει τα συμπεράσματα, ε, την ε, υλοποίηση μια συμφωνία, ε, την έχει αναβάλει για την επόμενη θητεία. Γι' αυτό και είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει και ο χρόνο πιέζει και σε αυτή την αβέβαιη περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έδινε ένα πολύ κακό αρνητικό μήνυμα αν δεν κατάφερε να καταλήξει συμφωνία πριν τα τέλη του έτου, ώστε να αποφύγουμε ένα επενδυτικό κενό όπω είχε συμβεί το 2014 όπως έχουμε υπενθυμίσει επανειλημμένως και στη διάσκεψη κορυφής των Δήμων και Περιφερειών ε, επήγει η λήψη συμφωνίας αλλά όχι μια συμφωνίας ε, τυχαία ή μια συμφωνία πάση θυσία. Χρειαζόμαστε μια καλή συμφωνία για τους Ευρωπαίους. Και εδώ θα ήθελα να σας δώσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε Αρτουή. Monsieur le Président, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, επιτρέψτε να σας πω πόσο είμαι ικανοποιημένος που μοιράζομαι αυτή τη στιγμή μαζί σας για να μιλήσω σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικό μας πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χαιρετίζω εσάς εκπροσώπους των περιφερειών, εκπροσωπείτε την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών χωρών, εσείς είσαστε σε, πραγματι... σε επαφή με την πραγματικότητα εσείς ακούτε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών τους αφουγκράζεστε λοιπόν διαρωτώ με κατά πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει στους Ευρωπαίους όταν το σκέφτομαι αυτό λέω στον εαυτό μου ότι είσαστε εκείνοι και εκείνες που επειδή είσαστε κοντά κοντά στους πολίτες και κοντά στις περιοχές αυτές είστε στην καλύτερη θέση εσείς για να ακούσετε τις προσδοκίες τους και να διαβιβάσετε τα μηνύματα. Πράγματι, αντιμετωπίζει δυσκολίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσκολίες όσον αφορά το να μιλήσει, να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους. Να σας πω ότι οι σχέσεις που διατηρούμε μεταξύ Επιτροπής Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την δική σας επιτροπή, την επιφορτισμένη με την εδαφική συνοχή και τον προϋπολογισμό, αυτές οι σχέσεις είναι έξοχες, εξαιρετικές. Έγινε κοινή προσπάθεια επί σειρά μηνών και δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω την πρόεδρο της Επιτροπής σας, την κυρία Μπουντινό, Θέλω να υπογραμμίσω σε ποιο βαθμό οι τοποθετήσει τη Επιτροπή Προπολογισμών και οι προσανατολισμοί τη Επιτροπή Προπολογισμών συντονίζονται με τι ανησυχίε που εξεφράστησαν από την Επιτροπή τη οποία ε, ηγείται. Προεδρεύω τη Επιτροπή Προπολογισμών και πράγματι, κύριε Πρόεδρε, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι μέτριο, μετριοπαθή. 1% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντο. Αν συγκρίνουμε αυτόν τον προπολογισμό με τον προπολογισμό των διαφόρων χωρών, είμαστε στο 45 με 50% του ΑΕΠ εκεί. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι 1%. Και τι κάνουμε εμείς με αυτό τον προπολογισμό που είναι μόλις τα, λίγο παραπάνω από τα δύο τρίτα που ε, τα δύο τρίτα πηγαίνουν στον στην κοινή αγροτική πολιτική και στο Ταμείο Πολιτικής Συνοχής στα Ταμεία Συνοχής ε, έχουν επιφανή θέση λοιπόν οι περιφέρειες ε, και η τοπική αυτοδιοίκηση στον προπολογισμό. Πώς χρηματοδοτείται προπολογισμό, χρηματοδοτείται από τους ιδίους ε, πόρους, τα τέλη που εισπάτονται σε εξωτερικά σύνορα, οι δασμοί που εισπάτονται σε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπογράφει ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, λιώνουν αυτά τα εισοδήματα σαν το χιόνι στον ήλιο ε, ανάλογα με τις ε, συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών και καρτούν και 20% οι χώρε για τον εαυτό του και αυτό που απομένει για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από του δασμού είναι μόλι 10%. Το 90% που προέρχεται, τα κράτη-μέλη προέρχεται. Ανάλογα με τον σχετικό του πλούτο. Εφόσον λέγεται ότι η κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής επιστρέφουν τους πόρους στα κράτη-μέλη, κάθε χρόνο έχουμε κάνει μια σύγκριση σχέση με αυτά που καταβάλει κάθε κράτος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και σε αυτά που δέχεται η χώρα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Λοιπόν, υπάρχουν οι χώρες εκείνες που πληρώνουν περισσότερα από αυτά που εισπράττουν και οι χώρες που αντίθετα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από αυτά που συνεισφέρουν. Και αυτό γρήγορα ε, καταλήγει σε βαθμό μηδέν αλληλεγγύης. Για να βγούμε από αυτό το θέμα και την τυραννία της σωστής επιστροφής χρημάτων προσπαθούμε να βρούμε νέους ιδίους πόρους ε, θα ήταν νέοι φόροι ίσως που ίσως άμεσα ε, να ε, αποδίδονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό δεν θα, αύξα, θα αύξανε τους ιδίους πόρους μεν, αλλά όχι το συνολικό πλαίσιο του προπολογισμού, το συνολικό όγκο του προπολογισμού. Εφόσον πρόκειται για νέους φόρους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Ευρωπαίοι, φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να ε, δεχτούν ε, πολύ μεγάλη αύξηση των ε, φόρων. Λοιπόν, θα επηρεαστούν οι ίδιοι πόροι από τους φόρους, αλλά για να τονωθεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμός θα πρέπει οι εθνικοί φόροι που εισπράττονται για τον προπολογισμό του κράτους ή των, ε, της να μειωθούν αναλογικά. Ποιο είναι το όφελο των νέων ιδίων πόρων. Είναι ότι μειώνουν αυτοί οι πόροι τη συνεισφορά των κρατών μελών και συνεπώ να βαρύνουν ε, αυτό το θέμα τη σωστή επιστροφή των χρημάτων. Λοιπόν, τη δίκαιη επιστροφή ίσως ε, θα είναι ένας φόρος των χρηματοδοτικών ε, συναλλαγών, μπορεί να είναι αυτός ο ίδιος πόρο. φόρος του άνθρακα στα εξωτερικά σύνορα, μπορεί να είναι αυτό, ένας φόρος όσον αφορά τα απόβλητα, ε, μια ποσότητα όσον αφορά τα κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, έχοντας επίγνωση ότι 28 χώρες είναι διαφορε... έχουν διαφορετική φορολογική βάση και κάθε εθνική νομοθεσία ε, έχει κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, ε, μειώσεις, κίνητρα φορολογικά που περιπλέκουν το εγχείρημα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση των νομοθεσιών, ώστε να καταλήξουμε σε ενιαία φορολογική βάση, αλλά ε, ένα τμήμα του, της φορολόγησης από τα κέντρα των επιχειρήσεων θα πρέπει απευθείας να καταβάλλεται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και όσο μας αφορά εδώ στο Κοινοβούλιο ε, συσχετίσαμε στενά τη συνεισφορά μας στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τη δημιουργία των νέων ε, ιδίων πόρων. Αυτό για να μειώσουμε τον αντίκτυπο ε, του αιτήματο για τη δίκαιη επιστροφή των συνεισφορών. Ε, αυτό είναι ένα εγχείρημα περίπλοκο στο οποίο έχουμε επιδοθεί ε, ε, λάβαμε γνώση όπως και εσείς τις προσπάθειες που καταβάλει ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2018 περιμέναμε σημαντική πρόοδο πάνω σε αυτό ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τέλος του έτους του 2017 είχε αναφερθεί στο ποσοστό του 1,2 του ΑΕΠ και αυτό που μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 1,11 με ένα μικρό τεχνούργημα θέλετε, δηλαδή ότι συνάθρισε στον προπολογισμό, συνυπολόγισε στον ευρωπαϊκό προπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Άμυνας που μέχρι τώρα δεν εμφανιζόταν καθόλου. Εάν βγάλουμε αυτή την προσθήκη είμαστε σε μια αύξηση του 1,08 και όχι 1,20. Το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι αυτό δεν ήταν η επιθυμία του, διότι είχαμε καθορίσει 1,3 θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να είναι το όριο του επόμενου προπολογισμού στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 γνωρίζοντας ότι το εγχείρημα θα είναι περίπλοκο και θα περιπλακεί από ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Λέω ενδεχόμενη αποχώρηση, διότι εδώ και μερικές εβδομάδες μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έβγαινε, βλέπαμε θα έβγαινε ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως ε, θα, θα ξέρουμε τι θα γίνει με τι διαπραγματεύσει απόψε τι επόμενε ε, ώρες υπάρξει ε, παράταση του χρονικού ορίου και δεν ξέρουμε αυτή η παράταση του χρονικού ορίου για την η αποχώρηση ποια θα είναι. Λέγαμε ότι το 2019 δεν θα υπήρχαν πιστός πέρα από τις 31 Μαρτίου για τους Ευρωπαίους βουλευτές, ευρωβουλευτές και τους συνεργάτες τους αλλά ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει έναν διορθωτικό ε, προπολογισμό για μια περίοδο που δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Και μετά, στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να λάβουν υπόψη νέε ανησυχίε. Αλλάζει ο κόσμο. Η παγκοσμιοποίηση μα δημιουργεί προηγουμένου προκλήσει όσον αφορά την ασφάλεια, όσον αφορά την άμυνα, όσον αφορά την ε, μετανάστευση, ε, όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία ένα γίγαντα του Ευρωπαίου της ψηφιακής τεχνολογίας πείτε μου όλοι είναι Αμερικανοί Αμερικανικοί φορεί ή Κινέζικοί λοιπόν και κατάφεραν μάλιστα να δημιουργήσουν φορολογικά συστήματα αυτοί ώστε στην Ευρώπη να μην ε, πληρώνουν φόρο στην Ευρώπη αυτοί οι ψηφιακοί γίγαντες ε, σε αυτά τα θέματα λοιπόν αν θέλουμε αποτελεσματικότητα δεν μπορεί παρά είναι ε, ευρωπαϊκή όπως τα, ε, γι' αυτό θεσπίσαμε και κανονισμό για προστασία των προσωπικών δεδομένων ψηφιακών στοιχείων ή ένα μηχανισμό για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και των διάφορων παρεμφερών δικαιωμάτων συγγενών δικαιωμάτων η Ευρώπη, μόνο μέσω Ευρώπης να το πετύχουμε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ε, υπολείπεται των προσδοκιών. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε δικό μας όραμα, να ψηφίσουμε δικό μας όραμα για το επομενο πολιτες πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Ε, το ποσοστό 1,3% το ΕΠ θέλουμε, λαμβάνοντα υπόψη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα το επανεξετάσουμε ενδεχομένω αυτό. Και θέσαμε σαν αρχή ότι οι πόροι που διατίθεται στην κοινή αγροτική πολιτική δεν θα πρέπει να περικοπούν από το επίπεδο το παρόν. Θεωρήσαμε επίσης ότι οι πιστώσεις για την πολιτική συνοχής θα πρέπει να παραμείνουν στο παρόν επίπεδο. Ε, ενώ σε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δική της εκδοχή υπάρχουν κάποιες ε, περικοπές. Είπαμε ότι οι πιστώσει του έρασμου πρέπει τριπλασιαστούν, οι πιστώσει για την έρευνα πρέπει σημαντικά να αυξηθούν, να πρικοδοτηθούν πέρα από το παρόν επίπεδο τη έρευνα είναι αυτή που ετοιμάζει το μέλλον μας. ουσιαστικά εκεί που κάπως ενοχληθήκαμε στην προσπάθεια που καταβάλαμε ήταν ότι το να προσπαθήσουμε ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2028 χωρίς να ξέρουμε για ποια Ευρώπη μιλάμε και τι ε, περιμένουμε από την Ευρώπη. Θέλουμε να την κάνουμε παγκόσμια δύναμη και πώ μπορεί να πιστέψει να θα κάνουμε μια παγκόσμια δύναμη με έναν προπολογισμό το 1,3% που κατανέμεται κατά 2 τρίτα στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτό είναι το θεμελιώδε θέμα. Ε, δεν έχει. Ίσως να το ζήσετε στην επικράτειά σας, στην ε, τοπική σας περιοχή διότι εκπροσωπείτε την ποικιλομορφία των διαφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να το ζείτε αυτό. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, να σας πω ότι δεν μπορούμε να τον προωθήσουμε, έχουμε πρόβλημα. Ε, εάν τελικά οδηγήσει σε μια αύξηση των δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι τα κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, δηλαδή ε, ε, οι δράσει όσον αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε που σήμερα εξασφαλίζονται από τα κράτη-μέλη. Αλλά λόγω της παγκοσμιοποίησης δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές υπηρεσίες όπως απαιτείται στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, Φερρυπίν, της μετανάστευσης, στον τομέα της προστασίας από την αλλαγή του κλίματος, για το περιβάλλον, ε, στον τομέα το ψηφιακό, ε, στο το εθνικό επίπεδο είναι το κατάλληλο επίπεδο. Εάν θεωρήσουμε ότι η δράση θα είναι αποτελεσματικότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιο αποτελεσματική από ότι στο επίπεδο κρατικό η πιστώσει στον οποίο η αποτελεσματικότητα δεν είναι στο κατάλληλο επίπεδο, μήπω θα μπορούν να βγουν από τον εθνικό προπολογισμό και τα χρήματα αυτά να μπουν στον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Είναι ένας μηχανισμός ε, που έχει ε, όπως γίνεται ε, γι' αυτό όπως όταν ζητάμε στις κοινότητες να ομαδοποιηθούν παρόμοια προσέγγιση και να δώσουν αρμοδιότητες στο πιο ομαδικό φορέα και το εισόδημα. Ε, θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό, αν θέλουμε λοιπόν η Ευρώπη να γίνει παγκόσμια δύναμη, είναι ένα θέμα προ συζήτηση. Είναι και διάφορες γεωπολιτικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η πολυμερής προσέγγιση όπως εφαρμόστηκε μέχρι τώρα ίσως ε, δεν αρκεί και ίσως ε, τα Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ρωσία, οι χώρες ήπειροι, η Ινδία, ίσως αύριο η Βραζιλία θα έχουν την τάση να μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους. Αν δεν ομαδοποιούν, δεν ενωθούν οι Ευρωπαίοι, ίσως να υποστούν την επιρροή και ίσως την κυριαρχία αυτών των χωρών που είναι ήπειροι ε, ε, ε, μέσω των οικονομικών και των μεγάλων ψηφιακών πολυεθνικών. Πρέπει να σκεφτούμε ποια θα πρέπει να είναι η Ευρώπη. Μια Ευρώπη που ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα προετοιμασία του μέλλοντο, του μέλλοντο των παιδιών μα. Μια Ευρώπη που μα προστατεύει. Μια Ευρώπη η οποία διακηρύσει την φιλοδοξία της να είναι μια παγκόσμια δύναμη η ισχύς όμως είναι στις περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο, ιδίω κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κάποιε σκέψει, γενικέ σκέψει που ήθελα να σα γνωστοποιήσω για να σα πω που βρισκόμαστε, υπογραμμίζοντα εκ νέου σε ποιο σημείο οι σχέσει μεταξύ τη Επιτροπή σα της Επιχωτισμένης για τις ε, περιφέρειες του προπολογισμού και της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σχέσεις εμπιστοσύνης. Ε, είναι σχέσεις αμοιβαίας συνδρομής, συνεργασίας, κοινής προσπάθειας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω διότι η μαρτυρία σας ε, ε για αυτά που είσαστε μάρτυρες αυτών που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, αυτούς τους τελευταίους μήνες από το 2016. Οι σχέσεις είναι στενές μεταξύ συνεισηγητών που προετοίμασαν τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με το Ευρωκοινοβούλιο. Μεταξύ της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου είναι πολύ καλές οι σχέσεις. Σας ευχαριστώ και εύχομαι αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθούν έτσι περαιτέρω προ κοινόν όφελο και όφελο των Ευρωπαίων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτήν την ε, κατάσταση πραγμάτων που μας περιγράψατε. Πολύ καλή παρουσίαση για την εισαγωγή του θέματος αυτού και σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για τη σημασία των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε για τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ιζαμπέλ Μπουντινού, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ΚΟΤΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Ζωάν Αρτσουή, τον πρόεδρο της Επιτροπής Προλογισμού του Κοινοβουλίου για αυτά που είπε για τη θαυμάσια συνεργασία μας. Και θα επανέλθω Όντω υπήρξε καρπο, καρποφόρα, αγαπητοί συνάδελφοι τη Επιτροπή Περιφερειών, και εγώ συμμερίζομαι την αισιοδοξία του τίτλου τη συζήτησή μα για έναν μελλοντικό προβλημό τη Ένωση που να ανταποκρίνεται στι φιλοδοξίε μα. Αλλά ακόμη δεν το έχουμε επιτύχει. Ο προπολογισμό, δυστυχώ, σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα ανταποκρίνεται στι φιλοδοξίε που εμεί, ω Επιτροπή Περιφερειών και όπω είπατε και εσεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιθυμούσατε για την Ευρώπη. Η Επιτροπή μας εκφράστηκε επανειλημμένα για τον προπολογισμό. Ιδιαίτερα μέσω τριών εκθέσεων που εγκρίναμε τους τελευταίους μήνες. Είχαμε αυτή για τους ίδιους πόρους, την οποία παρουσίασα εγώ και δεν θα επανέλθω, την περιέγραψε πολύ καλά και ο ε, Ζωάννα Ναχτούι, ε, την έκθεση επίσης του Μαρέκ Βοσνιάκ για το κείμενο θεωρητικής αναζήτησης για, ε, για την χρηματοδότηση του μέλλοντος τη Ευρώπης και την έκθεση επίση για του μελλοντικού προπολογισμού. Βεβαίω, η Επιτροπή Περιφερειών, όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελε τα κράτη-μέλη να ανεβάσουν στο 1,3% του ΑΕΠ ε, την συνεισφορά του. Αλλά, όπω υπόθηκε, από ό,τι φαίνεται, και πάλι θα καταλήξουμε στο 1,08 περίπου. Θα είναι ακριβώς η πρόταση της Κομισιόν που μετά τις συζητήσεις συνήθως ε, περικόπτεται στο Συμβούλιο. Όλα αυτά δεν θα ήταν τόσο δραματικά εάν το τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν εξαρτιόταν, όπω υπόθηκε, κατά πάνω 50% από τι εθνικέ συνεισφορέ. Και δυστυχώ κάποιε κυβερνήσει είναι αρκετά παρανοϊκέ. Από τη μία λένε ότι θέλουν περισσότερη ενοποίηση, περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη φιλοδοξία, αλλά δεν πληρώνουν για όλα αυτά. Και επιμένουν σε αυτή την τυραννία της ε, δίκαιης επιστροφής ή επιδιώκουν πάντα εκπτώσεις στη συνεισφορά τους. Επανερχόμεθα στο 88 όπου θα θέλαμε να επανέλθουμε στο 88 όταν οι εθνικές συνεισφορές ήταν μόνο 11%. Τότε ήταν ευκολότερες διαπραγματεύσεις, συντομότερες για τον ε, καθορισμό του προπολογισμού. Με νέους ίδιους πόρους θα είχαμε ένα νέο περιθώριο ελιγμών και θα μπορούσαμε επιτέλους να κάνουμε και έναν μακρόπνο σχεδιασμό για να είμαστε πραγματικά σε θέση να επηρεάσουμε το μέλλον μας. Να μην το εφιστάμεθα απλώ, να μην αποφασίζεται αλλού στον κόσμο. Όπως είπατε, με αυτά τα κράτη υπήρους που μας κοιτάνε και γλύφουν τα χίλια τους. Θέλουν να μας καταπιούν. Βεβαίω θέλουμε ίδιου πόρου. Ε, ω Επιτροπή Περιφερειών είπα ότι υπάρχουν διάφορε για τι μεγάλε ψηφιακέ επιχειρήσει, για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, για τα πλαστικά, για το δεξιό του άνθρακο. Αν και δεν θα θέλαμε να έχουμε φόρο επί προϊόντων, τον οποίο θα θέλαμε να σταματήσουμε την παραγωγή. Επίση, ω τοπικέ αρχέ, λέμε ότι είναι επίγον να υπάρξει σύμφωνα συμφωνία για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτω ώστε να εγγυθούμε την έγκριση των προγραμμάτων τη Ένωση εγκαίρω να μην ε, ε, στερέψουν τα διαθροτικά ταμεία, κάτι που θα έχει για τους δικαιούχους δραματικές επιπτώσεις. Τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο προχωρούν επί του κανονισμού, αλλά για τις συνολικές χρηματοδοτήσεις δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι πολίτες υποφέρουν από αυτή την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα. Λέγεται ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει πριν από τη Γερμανική Προεδρία, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 2020. Αυτό θα ήταν τεράστια καθυστέρηση. Το Συμβούλιο βεβαίω έχει εγκρίνει μερικέ συμφωνίε για το περιεχόμενο των νομοθετικών πρωτοβουλειών για το μηχανισμό τη διασύνδεση, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έρασμο, την ψηφιακή Ευρώπη, τη δημιουργική Ευρώπη, την άμυνα, την αλληλεγγύη. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα. Αλλά η ουσία του θέματος είναι αυτός καθεαυτός ο προπολισμός. Αυτός θα μας δώσει τα μέσα για την άσκηση των πολιτικών μας. Και εδώ ακόμη Περιμένουμε και ανησυχούμε πολύ γιατί τη το στο Συμβούλιο. Διαπραγματεύονται με τρόπο που δεν μα ικανοποιεί. Η Αυστριακή Προεδρία και τώρα η Ρουμανική Προεδρία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι διαφανεί οι διαπραγματεύσει. Δημιουργούσαν ένα πλαίσιο για τα περίφημα κουτιά διαπραγματεύσεων. Η Ρουμανική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε για να προχωρήσει. Με καρδιά. Αλλά έχουμε διάφορε μονομερεί αποφάσει που αφήνουν κατά μέρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα του συμπολίτε μα. Για άλλη μια φορά φοβάμαι ότι αυτέ οι διαπραγματεύσει μπορεί να καταλήξουν στην αρχή τη δίκαιη επιστροφή. Άρα στην ουσία λιγότεροι πόροι. 1% αρκεί για να ενισχύσουμε τη θέση μα στον κόσμο. Μα γελάνε στι ΗΠΑ και στην Κίνα όταν τα ακούν αυτά. Εμεί ω Επιτροπή Περιφερειών είμαστε κατά τη πτώση τη χρηματοδότηση τη πολιτική συνοχή και τη γεωργίας και τη ανάπτυξη ανάπτυξης της υπαίθρου. Δεν είναι δυνατόν να μην επιδείξει αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περιφέρειές τη, Γιατί ε, όλο και περισσότερο στρέφονται προς ε, τα διάφορα ταμεία και όχι προς επιδοτήσεις, τα διάφορα δηλαδή χρηματοδοτικά μέσα. Θέλουμε μια δίκαιη εφαρμογή της πολιτική συνοχή που να μην αφήνει κανένα στο περιθώριο. Η αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο εξαρτάται από αυτό. Το είπαμε. Και εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλή θέση. Ευχαριστώ τον κύριο Ζων Ατουί και τους εισηγητές Ζαμπέλ Τονάμα, Όλμπρικτ Ζεραντοπρέ, Γιανού Λεβαντόφσκι και γενικότερα την Επιτροπή Προπολογισμών που έκανε μια θαυμάσια εργασία σε συνεργασία με εμά. Τι χαιρετίζω. Είναι πρώτη φορά που τα δύο θεσμικά όργανα ανέπτυξαν τέτοιο βαθμό συνεργασία για την πολιτική συνοχή είχαμε 560 τροπολογίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προέκυψαν από τα δικά μας κείμενα εδώ. Και μπορούμε πραγματικά να είμαστε συλλογικά περήφανοι για τον απολογισμό αυτής της συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων. Το είπαμε επίσης και με την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. Σήμερα το πρωί σημειώσαμε και την θαυμάσια συνεργασία που είχαμε και προσπαθήσαμε να θέσουμε και κάποια ορόσημα για το επόμενο κοινοβούλιο για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Μέσω τέτοιου διαλόγου, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων και των περιφερειών που εκπροσωπούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ευρώπη που χρειάζονται οι πολίτες μας. Πρέπει η νομοθετική διαδικασία να είναι σε στενή σχέση με τις τοπικές δυναμικές, τις ε, περιφερειακές ιδιορυθμίες την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Επαναλαμβάνω, η πολιτική συνοχή δεν είναι παλιά κλασική πολιτική αρτηριοσκληρωμένη. Είναι μια πολιτική για όλους που βασίζεται σε σωστή τοπική διακυβέρνηση, σε γνώση της τοπικής πραγματικότητας. Θέλουμε οι δικές μας δομές που είναι στην πρώτη γραμμή τη καινοτομία και τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασία και ενό καλύτερου περιβάλλοντο, όλοι αυτοί μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μα και πρέπει να προστατευτούν από την κλιματική αλλαγή, τι οικονομικέ και κοινωνικέ αλλαγέ που θα μπορούσαν να τι ε, αποδυναμώσουν αν δεν υπάρχει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπουντίνο και πριν ξεκινήσω τη συζήτηση, θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο Αρτουή. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω τις παρατηρήσεις μου και να απαντήσω σε κάποια σχόλια της κυρίας Μπουτινό σε ό,τι αφορά την εκπόνηση του μελλοντικού πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε το πλαίσιο καθ' αυτό που προβλέπει για κάθε πρόγραμμα ένα ύψος πιστώσεων και αυτό βρίσκεται στα χέρια του Συμβουλίου που πρέπει να αποφασίσει με ομοφωνία. Για το ύψος των πιστώσεων, η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζεται σε μία αποδοχή, μία απόρριψη. Μπορεί να πει μόνο ναι ή όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν δίνεται να τροποποιήσει τη θέση του Συμβουλίου. Αλλά οι προβλεπόμενες πιστώσεις για κάθε δημοσιονομική γραμμή και για πρώτη φορά στο έγγραφο που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλάβαμε τον κίνδυνο να προτείνουμε εμεί ε, ύψο πιστώσεων. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου και αυτό το κάναμε για να ασκήσουμε κάποια πίεση στο Συμβούλιο. Αλλά από τη στιγμή που έχουν εγγραφεί οι πιστώσει ε, στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι να φτάσουν επί τόπου, χρειάζονται διάβλη και οι διάβλη είναι τα προγράμματα. Και τα προγράμματα διέπονται από κανονισμού. Και οι κανονισμοί αυτοί εμπίπτουν στη διαδικασία της συναπόφασης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό όμως που μας προβληματίζει και μας ανησυχεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι κάποιες κυβερνήσεις θέτουν ως όρο για την ε, έγκριση τη συμφωνία του στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το γεγονό ότι θα πρέπει να δεχτούμε την ΑΒ διάταξη στα προγράμματα. Ενώ το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προποθέτει ομοφωνία για την έγκρισή του. Αν λοιπόν το Συμβούλιο αρχίζει και προεξοφλεί κάποια τμήματα της σύνταξη των προγραμμάτων, ο ρόλος του, του Κοινοβουλίου στη συναπόφαση συρρυκνώνεται. Και για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο, εδώ και μήνες προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Και ε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, αρμόδιο είναι το ΕΚΟΦΗΝ. Αλλά για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και δεν είναι οι ίδιοι υπουργοί στα δύο συμβούλια. Και η συμφωνία στο Συμβούλιο θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα. Πριν από ένα μήνα μόλις ε, είχα πάει με τους συνεισηγητές που αναφέρατε ε, μετέβη στο Βουκουρέστι για άτυπο Συμβούλιο Υπουργών προκειμένου να ασκήσουμε πιέσεις στους υπουργούς για να μην ε, καθυστερήσουμε πολύ στη λήψη των αποφάσεων και να μην εγκριθεί καθυστερημένα ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στα τέλη του 2019 και το 2020 γιατί αν εγκριθούν καθυστερημένα τα προγράμματα και εσείς επί τόπου θα έχετε προβλήματα στην εφαρμογή τους και θυμάμαι τι έγινε το 2014 στα τέλη του 2013 εθετήθηκε το τότε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και είχαμε περίπου 25 ε, δις ε, καθυστερούμενες πληρωμές και το 2015 το ίδιο και από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν δυσαρεστήθηκαν γιατί είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται οι απλήρωτοι λογαριασμοί στα τέλη του 2013 και μάλιστα δεν μπορούσε να του εξοφλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτού του λογαριασμού. Γιατί έχουμε αφενός την ανάληψη υποχρεώσεων και αφετέρου τι πληρωμέ. Και υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό έχουμε τα υπόλοιπα προ εκαθάριση. Δηλαδή τι υποχρεώσει που αναλάβαμε δεν εξοφλήσαμε. 295 δις είναι το ύψος των υπολείπων προς εκαθάριση. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια από τον ίδιο τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ετήσιο. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα το 2020 και 2021 θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο που αντιμετωπίσαμε το 2014 και 2015. Δηλαδή μία πληθώρα ανεξόφλητων λογαριασμών χωρίς να έχουμε πιστώσεις πληρωμών για να τους εκαθαρίσουμε. Ε, μακάρι να είχαμε συμφωνία πριν τις ευρωεκλογέ. Αλλά από την άλλη ποιος μπορεί να πάει σε ευρωεκλογέ λέγοντας όποιο και να ψηφίσετε ο προϋπολογισμός ήδη έχει καθοριστεί μέχρι το 2027. Καταλαβαίνετε τι εννοώ κύριε Πρόεδρε. Οπότε υπάρχει όντως θέμα προς συζήτηση στην προεκλογική εκστρατεία που ξεκινά για τις ευρωεκλογέ. Και δεν ξέρω ποιες θα είναι τελικά οι προθεσμίες γιατί από τι αρχέ ε, Ιουλίου θα αρχίσει να συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στι αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε και Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ο Επίτροπος ε, που ετοίμασε το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Θα μπορέσει μέχρι τότε το Συμβούλιο να συμφωνήσει. Πολύ αμφιβάλλω. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα ο διάδοχος του Επιτρόπου Έτιγκερ θα αναλάβει τη διεκπαιρέωση της συμφωνίας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τα επιμέρους προγράμματα. Κυρία Πουντινό, όπως είπατε, ο προπολογισμό ε, δεν ανταπεξέρχεται στις ε, φιλοδοξίες μας και στις επιθυμίες μας. Αλλά το θέμα είναι ε, ότι βρίσκεται στα χέρια των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και αν θέλουμε έναν πιο γεμάτο προπολογισμό πιο σημαντικό, θα πρέπει η συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη για την Ευρώπη που επιθυμούμε, για το τι προσδοκούμε από την Ευρώπη. Γιατί πολύ συχνά ακούω επικρίσει μορφέ για την Ευρώπη που την κατηγορούν ότι δεν κάνει αυτά που την εμποδίζουν τα κράτη-μέλη ουσιαστικά να πραγματοποιήσει. Δεν φταίει η Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη είναι ανένδοτα. Γι' αυτό έχουμε μείνει στο 1% συμμετοχή του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματο. Η μόνη αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εμπορική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού η νομισματική πολιτική για τις χώρες της Ευρωζώνης και η προστασία των αλλιευτικών πόρων. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα σήμερα, ίσως δημιουργήσει στο μέλλον σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θα έχουμε ίσως πρόβλημα στις αλλιευτικές ζώνες, στα αλλιευτικά πεδία. Εσείς είστε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, είστε η πρώτη επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε φροντίστε όλα αυτά τα θέματα που είναι ουσιώδη για το μέλλον μας γιατί τα μέσα που θα έχουμε για να, να προστατευτούμε γιατί περιμένουμε από την Ευρώπη προστασία, ασφάλεια από πολλές απόψεις θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να λάβουν μέρος στη συζήτηση γιατί αν αφήσουμε τη συζήτηση μόνο σε επίπεδο κρατών μελών και δεν την κάνουν κτήμα του οι πολίτε, βλέπετε τι κατάληξη έχουμε κάθε φορά όταν μένουν τα, χέρ, τα πράγματα στα χέρια μόνο των κρατών μελών, των κυβερνήσεων. Πάντως όλοι σα είστε σε θέση να επικοινωνήσετε με σοφία και σύνεση στις περιφερειές σας και στους δήμους σας και ίσως εσείς καταφέρετε να προωθήσετε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις απαραίτητες ε, δημοσιονομικές συνέπειες. Ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε, θα μπούμε σε ανοιχτή συζήτηση, θα ακολουθήσουμε δύο στάδια. Να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές, δύο λεπτά ο καθένας. Μετά από το ζητήσω από τον κύριο Πρόεδρο να μιλήσει και πάλι. Μετά θα έχουμε 12 που θα παρέμβουν και θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και ο καθένας θα έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό. Από τους εισηγητές ξεκινάμε. Η κυρία Μαρίνη έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουν εισηγήτρια μαζί με τη συνάδελφο Σνάιντερ για τον κανονισμό για τις ε, κοινέ αυτές ε, διατάξεις και ομόφωνα υποστηρίχθηκε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Να εκφράσω εν συντομία σε δύο λεπτά κάποιες σκέψεις συνδέονται με μια εντολή που έδωσε η Επιτροπή των Περιφερειών στην τοποθέτησή μα που εκφράστηκε προ το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών είπε ότι η ποικιλομορφία των πόλεων και των περιφερειών είναι ένα στοιχείο ισχυρό. Καθορίζει την ταυτότητα και είναι η οικονομική και κοινωνική ισχύ τη Ευρώπη. Πρέπει να φροντίσουμε αυτή η ποικιλομορφία να μην ε, οδηγήσει σε αποστάσεις που θα δημιουργηθούν και διαφορές στην Ευρώπη. Η συζητήση του προπολογισμού εμά τη πόλη και τη περιφέρεια τη Ευρώπη, η πολιτική συνοχή και η προπτική τη πολιτική συνοχή παραμένουν θεμελιώδη στοιχεία. Όχι μόνο για το ρόλο μα ω τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι από αυτή την πολιτική εξαρτώνται πολλέ στατικέ επενδύσει ένα απτό όραμα της Ευρώπης για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για τις κοινότητές μας. Κάναμε σημαντικό έργο μαζί με τη Συμμαχία για τη Συνοχή όσον αφορά τις αρχικές προπτικές του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου οι περικοπές ίσως ήταν λιγότερες από αυτές που κινδυνεύαμε να έχουμε. Εκτιμήσαμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είχε ε, συνετάχθη με τις θέσεις μας. Όμως ανησυχούμε και θέλω να το καταλάβει και ο πρόεδρος αυτό. Διότι όσο πιο είναι πιο δύσκολη η συνεργασία με το Συμβούλιο. Ανησυχούμε όχι μόνο για την ε, ποσότητα, το ύψος του προπολογισμού, αλλά ίσως τελικά αυτή η πολιτική καταλήξει συμφωνία μεταξύ Βρυξελών και, και πρωτευουσών, με τις εθνικές κυβερνήσεις. Αντί η πολιτική να δίνει δύναμη στην τοπική αυτοδίκηση ε, και να οδηγεί σε συνεργασία και στην εφαρμογή τη αρχή επικουρικότητα. Το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο χρειαζόμαστε με σύγκληση. Το είδαμε στι κοινέ αυτέ διατάξει προσεγγίσεις. Χρειαζόμαστε σύγκληση Επιτροπή Περιφερειών και Ευρωκοινοβουλίου και έτσι αυτή η πολιτική να παραμείνει θεμελιώδης για τις κοινότητες, της πόλης και της ε, περιφέρειες. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ιόγκρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο. Σαν εισηγητής για την κοινή αγροτική πολιτική εκφράζω την ικανοποίησή μου και μπορώ να σας πω ότι έμβεντεύε και αγκρί στο Κοινοβούλιο ε, ενέκριναν διάφορες προτάσεις που κάναμε μέσω της γνωμοδοτήσεως και το οφείλουμε στην παρουσίαση της νομοδοτήσης Επιτροπής των Περιφερειών σε δύο κοινοβουλευτικές ακροάσεις. Συνεχώς υπήρξε συνεργασία με τους διάφορους ηγητές των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Υπήρξε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο Υπήρξαν πολλέ συναντήσει, το χαιρετίζω αυτό. Υπευλήθησαν συμβαστικέ τροπολογίε και λάβονται υπόψη οι απόψει μα. Όπω και εμεί και το Κοινοβούλιο θέλει να παραμείνει ο προπολογισμό του ΚΑΠ και να υπάρχουν περιορισμένε μεταφορέ στο δεύτερο προ τον πρώτο πυλώνα. Και για την κοινή οργάνωση τη αγορά υιοθετήθηκαν οι διάφορε διατάξει με Μητροπή Γεωργία. Επίση, ο ρόλο των περιφερειών στη διαχείριση και εφαρμογή τη ΚΑΠ ελήφθησαν υπόψη συμβαστικέ τροπολογίε του κανονισμού σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια που υθετήθηκε στι 2 Απριλίου. Αυτή η υποστήριξη του Κοινοβουλίου είναι σημαντική. Όταν τα κράτη-μέλη θέλουν ξανά κεντρική διαχείριση τη κοινή αγροτική πολιτική. Τα κράτη-μέλη για την ώρα δεν, δεν εισακούν τα διαβήματά μα. Στι 13 Μαου, στη διάσκεψη υψηλού επίπεδου που διοργανώνεται από τη Ρωμανία Γερμανική Προεδρία για την ΚΑΠ θα πρέπει να τα επαναλάβουμε αυτά. Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και όλε για να πείσουμε του ηγέτε των διαφόρων χωρών μα να λάβουμε καλύτερα υπόψη τη φωνή των περιφερειών στην υλοποίηση και εφαρμογή τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που είναι ε, κάτι απαραίτητο για την ανάπτυξη των περιφερειών. Λείπει ε, στην επιτοπή, Γεωργία, λείπει φιλοδοξία στον αφορά τη σωστή κατανομή των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά των τρόπων τη βιώσιμη παραγωγή. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα προ μια ΚΑΠ που είναι βιώσιμη, δίκαιη και αλληλεγγύη που ζητά η Επιτροπή των Περιφερειών να λάβουμε υπόψη διάφορε στοιχείε κλιματικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ. Συνεχίσω την εργασία μου απευθυνόμενο προ το παρόν και μελλοντικό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ζητήσουμε σημαντικά κονδύλια να αφαιρθούν ε, για τη σωστή κατανομή και οι στόχοι ευρωπαϊκοί προσμετρήσιμοι ε, μέσω εθνικών στρατηγικών σχεδίων να συμπεριφθούν στον κανονισμό για να αποφευχθούν τον ανταγωνισμού μεταξύ κρατών μελών και επιτέλους να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά και του κλίματος. Και τώρα, Κριστόφ Κλαβζού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ολοκληρώνεται η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας εκπροσωπείτε τους ε, συμπολίτες μας από την περιφέρειά μου. Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής σας ζωής για μια σωστή απάντηση, συλλογική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είμαι για το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη ε, που είναι από αυτούς που κέρδισαν σε αυτή τη ζήτηση. Ορισμένοι θέλουν ε, ακόμη περισσότερε πιστώσει για το ορίζον Ευρώπη. Και εγώ θα ήθελα, εάν ήταν απεριόριστα τα χρήματα. Αλλά το βασικό είναι να διατηρηθεί ο προπολογισμό τη κοινή γεωργικής πολιτική και τη πολιτική συνοχή. Μπορούμε βεβαίως να θέλουμε και καλύτερη λειτουργία της πολιτικής ε, έρευνας. Αλλά αν ήμουν ερευνητής θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το τι κάνει η Ευρώπη για την έρευνα, για την ανώτατη εκπαίδευση, για την νεότητα. Είναι κατακαιρματισμένες αυτές οι πολιτικές σήμερα και δεν φαίνεται ποια είναι η συνολική τους επίπτωση. Και δεύτερον, αν θέλαμε να έχουμε φιλόδοξο όραμα, θα έπρεπε να μπορούμε να συνδυάσουμε τα χρήματα του, προγράμμα, του προγράμματος έρευνα, προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και του προγράμματος ε, περιφερειακής συνοχής. Καταλήγοντας, Ακούγοντά σα, κύριε Πρόεδρε, ίσω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το εξή. Διότι πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα στην Ευρώπη ή πρέπει να δαπανίσουμε διαφορετικά, με διαφορετική κατανομή των πόρων μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι δεν επενδύουμε αρκετά για την έρευνα και ανάπτυξη, για την νεότητα, για, να, ε, για την οικολογική και ενεργειακή μετάβαση. Και τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι ζωτικά για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Θα χρειαστεί λοιπόν να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για περισσότερες επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος μας, ο Μάρκου Μάρκουλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κρίστοφερ Κλερζό. Πρέπει να είμαστε πιο ρηξικέλευθοι στην προσέγγιση μας. Πού είναι οι ανάγκη στην Ευρώπη, κυρίως στη νέα γνώση, την ε, ψηφιοποίηση και την ένταξη της έρευνας στην προσπάθεια επιτάχυνσης της καινοτομίας. και εκπροσωπώ την άποψη όχι μόνο της ομάδας μου αλλά και των άλλων συναδέλφων πιστεύω λέγοντας ότι χαιρόμεθα που το Κοινοβούλιο εστίασε εκεί που εστίασε και πρέπει να επιμείνουμε πρέπει να συνεργαστούμε όλο και στενότερα και εμείς όταν επιστρέφουμε στις περιφέρειες και στις πόλεις μας και μιλάμε με τους πολίτες μας και με τα πανεπιστήμια και τους οικονομικούς παράγοντες πρέπει να αποδείξουμε ότι ορισμένες επενδύσεις πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ζωτικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν το 1,3 και όχι μόνο αυτό το 1,0 δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά είναι ευθύνη όλων μας. Πρέπει να πείσουμε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις ότι αυτές είναι οι καλύτερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε. Η απόδοση των επενδύσεων αυτών είναι καταπληκτική ιδιαίτερα η χρήση της ψηφιοποίησης και μέσω της προώθησης του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Βεβαίως, πρέπει να στηρίξουμε τις, τις χρηματοδοτήσεις που έχουν επιτευχθεί γι' αυτό. Και αυτά λέγαμε και στη δική μας γνωμοδότηση. Ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Το δίκτυο των κόμβων ευρωπαϊκής ψηφιακής καινοτομίας είναι αναγκαίο παντού. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε περιφέρεια. Πρέπει να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δίκτυο αυτό. Όπου να συμμετέχουν ε, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσω αυτών των ε, ομήλων. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο ε, πόλο που να ανταγωνίζεται τους υπάρχοντες. Θέλουμε να τα συνδυάσουμε. Είναι πολύ καλό παράδειγμα η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας επιτρέπει να φτάσουμε στην κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίε μας. Έχουμε και μια παγκόσμια ευθύνη να αποδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο και να βοηθήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που είναι ενώπιόν μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ουλρικέ Χελό. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εισηγήτρια για το πρόγραμμα που θα είναι συνέχεια του Έρασμο ΣΥΝ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνωμοδότησή του στην ουσία υιοθέτησε με πολύ λίγες αλλαγές τη δική μας. Και εμείς λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν το πρόγραμμα που θα δεχθεί το σύν από τη μία να βοηθήσει τους μαθητευόμενους αλλά και την διαβίου κατάρτιση από το σχολείο μέχρι τους ηλικιωμένους και επίσης θέλουμε οι νέοι να μπορούν να έχουν εμπειρίες ε, πέρα από τη χώρα τους αναξάρτητα από τις δυνατότητες των γονέων τους και ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να απλουστευτεί και ε, θαραλέω αλλά και πονηρό ε, είναι αυτό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τριπλασιασμό των πορών, δηλαδή 140 δις. Εμείς προτείναμε μόνο 30. Το στηρίζω πολύ καλά αυτό. Ελπίζω και στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις να επιτύχουμε περισσότερα. Όντως να μπορούν περισσότερο να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και αυτό πιστεύω θα είναι προς το συμφέρον όλων μας, αλλά ιδιαίτερα προς το συμφέρον των νέων μας, κοριτσιών και αγοριών που θέλουμε να τους κερδίσουμε για την Ευρώπη, να έχουν μια σωστή ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η Μαρία Αντωνέτ Μοπεχτουή έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον κύριο Ζανάρτουη που είχε την καλοσύνη να έρθει για να συζητήσουμε. Είμαι η συγκεκριτήρια στην πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ε, στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό η Επιτροπή μείωσε κατά 12% τα κονδύλια για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνοχή ε, που είναι κάτι πολύ ορατό για τους πολίτες και τις τοπικούς και περιφερειακούς φορείς μέσω του προγράμματος Interreg που είναι πολύ καταξιωμένο πρόγραμμα γιατί επιτρέπει τη σύγκληση των πολιτών με τους ε, τοπικούς φορείς και έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία γιατί φέρνει και τους πολίτες πιο κοντά μεταξύ τους. Ε, στη γνωμοδότηση του Δεκεμβρίου του 2018 η Επιτροπή των Περιφερειών ε, ζήτησε τη διαφύλαξη των 10 δισεκατομμύριων ευρώ του ποσού για το, την πολιτική αυτή και 970 επιπλέον εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία. Τα αιτήματά μας τα διαβιβάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συντονισμένη συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Ρημό και την Επιτροπή Ρέγγι μας επέτρεψαν να συγκλίνουμε προς μια κοινή θέση και στις 28 Μαρτίου υιοθετήθηκαν αυτές οι προτάσεις μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα το πλαίσιο και ο μελλοντικό προπολογισμό του προγράμματο αυτού τη εδαφική συνεργασία βρίσκονται στο Συμβούλιο. Έχω δύο απορίε και περιμένω τα φώτα της εμπειρίας σας εδώ. Τι πολιτική κατά τη γνώμη σας ε, Ποιε πολιτικέ κατά τη γνώμη σα θα επηρεαστούν κυρίως ε, δημοσιονομικά από τις περικοπές και θεωρείτε ότι στο μέλλον ε, θα καταφέρουμε με τις ε, διαπραγματεύσεις να κρατήσουμε αρκετά υψηλά κονδύλια για την εδαφική συνεργασία που όπως σας είπα καλύπτουν τη διασυνοριακή συνεργασία τα κονδύλια αυτά, την διαπεριφερειακή συνεργασία και η Επιτροπή Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε και η ναυτιλιακή συνεργασία να παραμείνει στο διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, συνεργασία με τα υπερπόντια διαμερίσματα και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, με την διαπεριφερειακή συνεργασία Interreg Europe και τα διαπεριφερειακά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Αυτά, ευχαριστώ. Ακούσαμε όλους τους συζητητές για τον προϋπολογισμό και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στον πρόεδρο ε, Αρτουή για να απαντήσει. Θα ήθελα πρώτα να πω κύριε Πρόεδρε ότι όντω για αρκετά προγράμματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκρισταλώσει τη θέση του με απόφαση και τη Ολομέλεια. και είχαμε και κάποιου κάποιους διαλόγου, διαλόγους αλλά τα συμπεράσματα παρόλα αυτά όλων αυτών είναι προσωρινά γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη το ύψο των πιστώσεων και σε, όπως ε, γενικώ στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αν δεν συμφωνήσουμε για τα πάντα, δεν έχουμε συμφωνήσει για τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το έχετε κατά νου. Η κυρία Μαρίνη τόνισε την πολυμορφία των Δήμων και των Περιφερειών και ανέδειξε τη δυσκολία συνεργασίας με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την αμέριστη ελληνική μας. Και εμείς έχουμε προβλήματα στη συνεργασία μας με το Συμβούλιο. Και σε κάθε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προσπαθούμε πώς και πώς να ενημερωθούμε για το τι θα συμβεί ε, και να μπούμε σε αυτά τα κουτιά των διαπραγματεύσεων, αλλά κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έχουμε μια ενημέρωση των διαμυφθέντων για να, ενημερωθούμε για την πρόοδο που σημειώθηκε στο Συμβούλιο. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε διαπιστώσει σημαντική πρόοδο σαν να περιμέναμε κάποια μέρα να συναντηθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, να τους συγκαλέσει ε, σε ένα εξομολογητήριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να τους ε, ρωτήσει τι προσδοκούν και ως διαμαγείας να ε, υιοθετηθούν τα πάντα και να διευθετηθούν όλα. Δεν θα συμβαίνουν όμως ε, έτσι, δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα και ελπίζω η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρεμποδίσει ε, την υιοθέτηση των αποφάσεων κρυπτό και παραβίστο. η Ευρωπαϊκή, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό τη ΚΑΠ, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να εξο, εξισωθούν οι άμεσες ε, ενισχύσεις μέχρι τα τέλη του 2027 και το τέλος του ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Επίσης θα πρέπει να αναδειχθεί ο ρόλος των περιφερειών και μερικές φορές ε, στους κανονισμούς έχουμε περίπλοκες διατάξεις και μερικές φορές σε εθνικό επίπεδο έχουμε έναν κανονιστικό υπερθεματισμό αλλά ε, μερικές φορές υποπτευόμαστε για τέτοιο κανονικό υπερθεματισμό και τι περιφέρειες. Με παρεξηγείτε και μην παίρνετε στραβά, αλλά όλοι οι νομοθέτε είναι ύποπτοι για αύξηση της περιπλοκότητας της νομοθεσίας και η προσπάθεια κατάρτισης του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, με το χέρι μας στα τρέμει όπως έλεγε και ο Μότες και όταν εκπονούμε νομοθεσία. Ε, Κύριε Κλερζό, είμαστε αλληλέγγυοι και για τα θέματα της έρευνας και έχουμε προκήρυξη διαγωνισμών και τα πολύ καλά προγράμματα ε, δυστυχώς μόνο σε πολύ χαμηλό ποσοστό ικανοποιούνται 11% οπότε υπάρχει μεγάλη απογοήτευση ακόμη και είναι καλά τα προγράμματα και αξιόλογα είναι τόσο περίπλοκοι οι κανονισμοί που σε πολλές περιπτώσεις πρέπει κανείς να περάσει από ειδικευμένα γραφεία που ε, ε, λαμβάνουν τέλη επιτυχίας. Και μια και δεν είναι ευανάγνωστα τα προγράμματα όταν τα συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μερικές φορές ε, πρέπει οι δικαιούχοι να περνάνε μέσω εταιριών παροχής συμβουλών που χρεώνουν υπέρογκα τέλη επιτυχίας για να μην μιλήσω για τους ελέγχους εκ των προτέρων, εκ των υστέρων και μία σειρά ελέγχων που γίνονται στη διάρκεια των προγραμμάτων, όλες αυτές οι διαδικασίες αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους και δεν δίνουν την καλύτερη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο οι δαπάνες, γιατί το ύψος των δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη ε, συνολικά δεν μπορεί να αυξηθεί. Οπότε είναι καθήκον μας να λάβουμε γενναίες αποφάσεις, να μην αυξήσουμε τις δαπάνες και μερικές φορές κάποια κονδύλια που δεν αξιοποιούνται καλά σε εθνικό επίπεδο να τα μεταφέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δείξουμε την ευρωπαϊκή αξία, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έχουμε καθήκον μονίμως να αποδεικνύουμε ότι αν τα κονδύλια που έρχονται, προέρχονται κυρίως από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αν περνάν από τον κοινοτικό προπολογισμό θα πρέπει να έχουν μια ορατή προστιθέμενη αξία που δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ελληνική. Κύριε Πρώτε Αντιπρόεδρε, επιμείνατε στην ανάγκη συνεργασίας, στην ανάγκη να αφογκραστούμε τους πολίτες, επιμείνατε στην ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση σίγουρα είναι από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί θα διακυβεύσει ολόκληρους επαγγελματικού κλάδους. Χθες στο κτίριο Σαλμάνιχ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μια διάσκεψη ε, με θέμα το μέλλον της ε, απασχόλησης. Οπότε έχει μεγάλη σημασία η επαγγελματική κατάρτιση για να προετοιμάσουμε τα νέα ταλέντα και όχι μόνο ε, η, ανώτερη, η εκπαίδευση και ανώτατη εκπαίδευση. Η κυρία Μίλλερ μίλησε για το έρασμος και εδώ συμφωνούμε. Φυσικά είναι προς το συμφέρον μας να τριπλασιάσουμε τα κονδύλια του Εράσμους. Ήταν ε, 1,5 δις και το 2014 και το 2019 μόνο θα κινητοποιήσουμε 3 δις. Σχεδόν έχουμε διπλασιάσει τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Αν μέναμε στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2021 θα είχαμε κονδύλιο χαμηλότερο από το 2020. Γιατί σήμερα το έρασμος ε, καλύπτει μόνο τις μισές αιτήσει. Και αν δεν θέλουμε να περιοριστεί μόνο στους ε, φοιτητές και στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά θέλουμε να εκδημοκρατήσουμε το έρασμος και να επιτρέψουμε και στους μαθητευόμενους και στους ασκούμενους να υποφεληθούν από υποτροφίες ε, έρασμος, όχι μόνο για δύο εβδομάδες, αλλά για τουλάχιστον έξι μήνες εντατικά ε, σεμινάρια και να είναι λογικό να μπορεί να, ο μαθητευόμενος να μιλάει και άλλη γλώσσα πλέον της μητρικής του το Έρασμος πρόβλεψε τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τα κέντρα επαγγελματική κατάρτισης, τέτοιου είδους κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να βρίσκονται στην αιχμή των επιδόσεων. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την παιδεία και την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά έχουμε κάποιου μηχανισμού. Έχουμε την κινητικότητα μέσω του έρασμο, αλλά έχουμε και το μηχανισμό που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη. Με τα δύο αυτά ταμεία μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε επενδύσει ώστε αυτά τα κέντρα επαγγελματική κατάρτιση και κατάρτιση μαθητευομένων, μαθητευομένων ακόμη και σε χώρες που δεν υπάρχει τίποτα να εξασφαλίσουμε έξοδα χρηματοδότησης για να ε, εξυπηρετήσουμε μαθητευόμενους που προέρχονται από άλλες χώρες. Κυρία Μομπερσουή, θέσατε δύο ερωτήσεις, ε, Δύσκολα μπορώ να απαντήσω, διότι δεν γνωρίζω ποια είναι η θέση, θα είναι η θέση του Συμβουλίου στην τελική φάση. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το Κοινοβούλιο θυγραμμίζεται με εσά, διότι ζητήσαμε να διατηρηθούν οι πιστώσεις για τη συνοχή. Μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι ήταν λίγο αυθαίρετη η κατανομή των πιστώσεων συνοχή. Ήταν κάπω μια μαύρη τρύπα τη δημοκρατία που επικρατούσε εκεί. Το ελεκτικό συνέδριο συνέταξε έξοχη έκθεση που υπενθύμησε ποιε είναι οι παράμετροι που επέτρεψαν τις συμφωνίες του Δουβλίνου του 90 Σίγουρα υπάρχουν παράμετροι προσαρμογής για κάθε χώρα. Εμείς που μπορώ να πω που είμαστε υπεύθυνοι για τον όγκο να πούμε ναι ή όχι για το ποσό έχουμε αρμοδιότητα για τα προγράμματα διότι πρόκειται περί συναποφάσεως αλλά για αυτά τα θέματα που αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική ή τα ταμεία συνοχής είναι το Συμβούλιο που έχει τα πράγματα στα χέρια του και όπω έλεγε η κυρία Μαρίνη αν εσείς έχετε προβλήματα για να άμεσα να παίρνετε σε απαντήσεις που θέλετε από το Συμβούλιο, πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να ότι σας εισακούει το Κοινοβούλιο διότι παρά τις προσπάθειές μας έχουμε μεγάλο πρόβλημα ε, όσον αφορά να προβλέψουμε τι θα αποφασίσει αύριο το Συμβούλιο όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή τα διάφορα προγράμματα. Ιδού κύριε Πρόεδρε κάποιες απαντήσεις που θεωρώ ότι μπορούσα να δώσω. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε τώρα τη συζήτησή μας. Έχουμε 11 συμμετέχοντες που ζήτησαν να εγγραφούν στον κατάλογο των ομιλητών και θα κλείσω τώρα τον κατάλογο αυτόν. Σας επισημαίνω ότι χρόνος αγόρευσης είναι ένα λεπτό ανακεφαλή. Μίσιλ Ράις Βέρμαν, πρώτος ομιλητής, συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημαντική αυτή η συζήτηση. Είδαμε ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής των Περιφερειών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πολιτική συνοχής. παρακολούθησε τι εργασίε σαν εισηγητή, Υπήρχε έξοχη συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων. Υπάρχει σύγκληση απόψεων επί της ουσίας και η θέση του Κοινοβουλίου συμπίπτει με τη θέση της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτικής συνοχής στα σημερινά επίπεδα στο μέλλον υπάρχουν ισχυρές πιέσεις. Απειλείται αυτή η πολιτική αλλά σίγουρα η απειλή δεν προέρχεται από τα δικά μας θεσμικά όργανα, αλλά από τα κράτη-μέλη προέρχεται αυτή η απειλή. Όσον αφορά τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αποφάσεις για το InvestEU, για το Horizon Europe, λαμβάνονται αποφάσεις σαν να επιλέγονται θέματα από ένα ευχολόγιο και μετά ε, νομίζω τελικά θα παραμείνει τελευταία η πολιτική συνοχής και, τελικά τελευταίο θα είναι ε, αυτός που φτάνει στη γραμμή τερματισμού η πολιτική συνοχή. Πρέπει να σκίσουμε πιέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τηρηθούν οι συμφωνίε στην πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αναφέρω την αστική διάσταση πιο πολύ. Στην Ευρώπη όλο και περισσότεροι μένουν σε αστικά κέντρα. Ο ΣΑ υπολογίζει ότι το 2030 80% των πολιτών της Ευρώπης θα ζει σε πόλεις. Και δεν είναι μόνο πολύ μεγάλες πόλεις, είναι και πόλεις με έως 50.000 πληθυσμό. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν σωστό να λάβει περισσότερο αυτά, αυτή την αστική διάσταση στην πολιτική της. Ξέρω πόσο έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τα εκτιμώ, αλλά εφόσον συζητάμε το πι, Πρέπει να τονίσω ότι αυτή η διάσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη ακόμη σοβαρότερα. Αυτό αφορά τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγι, αλλά και τα ε, μέσα εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής που πρέπει να στραφούν προς τις πόλεις και το ορίζον 2020 που θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τις αστικές περιοχές. Η οργάνωση EuroCities απέτησε να υπάρχει ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να ασχολείται με θέματα πόλεων. Η Επιτροπή μας θα έπρεπε να προωθήσει περαιτέρω αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπρούνο Βράνικ, συνάδελφο, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει. Θα πρέπει όμως να εξορροπήσουμε τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Η πολιτική θα πρέπει να είναι παρκώς πρικοδοτημένη ώστε να εξισορροπήσει αυτές τις διαφορές. Και υπάρχει μεγάλη αλλαγή, ε, ανάγκη για μείωση των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη πολιτική συνοχής. Χαιρετίζω την πρόταση τη επιτροπή να γίνουν μεγαλύτερε επενδυτικέ προσπάθειε για, ε, για την νεολαία, του μετανάστε, ε, την έρευνα και εκεί θα πρέπει να πρωτοστατήσουν οι, Ευρωπαίοι, οι περιφερειακές αρχές αυτές τις επενδύσεις. Δεν θέλουμε να μειωθεί κατά 10% ο προπολογισμό τη πολιτική συνοχή, γιατί έτσι θα δικαιωθεί και το μέλλον τη πολιτική συνοχή. Και τέτοιε περικοπέ θα απειλήσουν σοβαρότατα την ίδια την πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπο ε, ε, που μεταφέρουμε κονδύλια της συνοχής σε κεντρικά προγράμματα δεν θα συμβάλλει στην εξορρόπηση των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η συρρήκνωση των κονδυλίων της συνοχής μας δημιουργεί την απορία για την επικουρικότητα γιατί η πολιτική συνοχή θα έχει μεγάλο ρόλο και στο επόμενο πι. Αλλά σήμερα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο την πολιτική συνοχή από ό,τι στο παρελθόν. Τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει ο στόχο να έχουν την εξορρόπηση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και των ευρωπαίων πολιτών. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε περικοπή κατά 10% των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Δυστυχώς έχει έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος αγορευσή σα, Ο κύριος Βάλτερ Νίγκο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τους στόχους μας. Ποιο είναι ο στόχο μας. Ε, να είναι η Ευρώπη ε, τόπος ασφαλούς διαβίωσης και τρόπος που θα επιτρέπει την ε, εκπλήρωση και την ανάπτυξη του ανθρώπου. Θα πρέπει να δούμε προτεραιότητες. Προτεραιότητες είναι η παιδεία, παιδεία που θα συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η καταπολέμηση της φτώχειας, η πρόσβαση όλων των πολιτών στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που θα στηρίζονται στη ψηφιοποίηση. Είμαι βέβαιος ότι ο κινητικός προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς τους στόχους και τις προτεραιότητες και να δημιουργήσει ούριο άνεμο για όλους αυτούς τους στόχους. Ο μελλοντικό κοινοτικό προπολογισμό θα πρέπει να αναδείξει και να στηρίξει όλες αυτές τις πολιτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Birgit Ευχαριστώ. Είμαι Υπουργό για Ευρωπαϊκέ Υποθέσει στη χώρα μου. Και θα ήθελα να στηρίξω αυτό το οποίο υπόθηκε. Ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση για την Κομισιόν και να μπορέσει να ανταποκριθεί στα μελλοντικά καθήκοντά της Ευρώπη. Ιδιαίτερα λόγω των επιπτώσεων του Brexit. Και επειδή Ήδη οι αρχοί κρατών κυβερνήσεων έχουν καθορίσει και νέε προτεραιότητε. Γι' αυτό είναι αναγκαίο τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του, να αυξηθεί ο προπολογισμό και για το Ερασμοσύν και για τα προγράμματα συνοχή. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Και επίση τονίζω ότι η Κομισιόν θα ε, πρέπει να έχει τους, δικός, τους δικούς της πόρους. Για παράδειγμα, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Κοινός στόχος πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικέ προκλήσεις. Γιατί εάν καθυστερήσει η έγκριση των προγραμμάτων συνοχής θα καθυστερήσει και η έγκριση της νέας γεωργικής πολιτικής για δύο-τρία χρόνια. Αυτά μας ανησυχούν ιδιαίτερα στη Γερμανία. Παρακαλώ να τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σίλικο Τούρκ. Συνάδελφος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την υποστήριξή μου στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αύξηση της ε, στήριξης του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη ε, των πόλεων και των ε, υπαίθρων και της υπαίθρου. Και τα κονδύλια αυτό των προγραμμάτων για, για το πρόγραμμα Urban, για το πρόγραμμα για τα αστικά κέντρα, για την εδαφική συνοχή και για τη δημιουργία ικανοτήτων στις ευρωπαϊκές πόλεις θα συμβάλλει στην πρόθεση της καινοτομίας και στις νέες προδιαγραφές στην κατασκευή κτηρίων στις πόλεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε φυσικά και τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων για να, ε, για να έχουμε ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και πολλοδομία και φυσικά να λαμβάνουμε υπόψη κοινωνικά, οικολογικά και ε, οικονομικά κριτήρια και τις αντίστοιχες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πίτερ Κάιζερ, ο συνάδελφος, έχει το λόγο. Οι προπολογισμοί είναι η πολιτική εκφρασμένη με νούμερα. Εκφράζει την πολιτική που θέλει ο καθένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μα θέλουν περισσότερη Ευρώπη. Θέλουν ε, προώθηση της περιφερειακής πολιτικής και δεν θέλουν καμία υπαναχώρηση στην πολιτική συνοχή. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τα κρατικά συμφέροντα με τα συμφέροντα των περιφερειών. Εδώ ήδη υπάρχουν διαφορές απόψεων και θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε το σωστό συμβιβασμό. Είναι σαφές ωστόσο ότι οι περικοπές στην πολιτική συνοχής, την περιφερειακή πολιτική, είναι η παναχώρηση για την Ευρώπη. Για τα έσοδα, να πω το εξή. Πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι για την φορολόγηση των ε, ψηφιακών γιγάντων και περισσότερο θάρρος για τη χρηματοδότηση για την ε, φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επιπλέον, τι έννοια έχει επίσης να ξανασκεφτούμε κάποια κριτήρια ε, ε, σύγκλησης που αναφέρονται στη συνθήκη του Μάστρεχτ. Ευχαριστώ. Ο έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα σε αυτά που μας κάνουν περισσότερο Ευρωπαίους. Κυρίως όσον αφορά την νεολαία, τον πολιτισμό και την πολιτική συνοχής για την νεολαία. Έχουμε την πιο φιλοευρωπαϊκή ε, γενιά στην ιστορία της Ευρώπης. Πρέπει να επενδύσουμε στο Erasmus Plus για τη μείωση της ανεργίας και άλλα προγράμματα για την νεολαία, για τον πολιτισμό η Ευρώπη αφορούσε πολύ ε, το σώμα και λίγο την ψυχή. Και τώρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα για την ψυχή της Ευρώπης. Δεν χρειαζόμαστε μόνο τα θεσμικά όργανα, χρειαζόμαστε όμως ε, τους πολίτες που είναι η ψυχή ε, της Ευρώπης και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τρίτον, η πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να είναι πολιτικός στόχος και όχι τεχνικός. Διότι το μέλλον μα, η Ευρώπη μα, εξαρτάται από την πολιτική συνοχή. Βλέπετε τα αποτελέσματα σε κάθε γωνιά τη Ευρώπη. Ανησυχώ πολύ για τη μείωση των πόρων για την πολιτική συνοχή, για την κεντρική διαδικασία και τη μείωση των ποσοστών συγχρηματοδότηση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ζούραικ Ντόμπλα. Ο συνάδελφο έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει πολλέ προκλήσει. Το Brexit, την ασφάλεια πολλά προβλήματα. Βασικό πυλών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όμω είναι η πολιτική συνοχή. Ξέρουμε ότι θα έχουμε μειωμένο προπολογισμό. Αυτό είναι μεγάλη πίεση για να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα χρήματα. Είναι τα εργαλεία που θα μα κάνει να χρησιμοποιήσουμε ευθεώ τα χρήματα είναι η ευελιξία. Η ευελιξία είναι ε, το, η λέξη κλειδί για την προσοχή. σαν πρόεδρο πιο ανεπτυγμένη περιοχή βλέπω μεγάλο αντίκτυπο για τη μεταφορά χρηματοδότηση μεταξύ κατηγοριών των περιφερειών και καλωσορίζω την Πρωθυπουργική Επιτροπή να αυξήσει την ευελιξία από 3 στα 15%. Χωρί αμφισβητώ ότι πρέπει υποστήριξη πρέπει να πηγαίνει σε λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ. Συμφωνώ με αυτό απολύτω, αλλά έχει νόημα χώρε να αποφασίζουν μόνε του πού πηγαίνουν τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Να τονίσω ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι μητροπολιτικέ περιοχέ που έχουν ειδικέ ανάγκε, κάτι που συνδέεται με κοινωνική ένταξη, περιβάλλον και μεταφορέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ομιλητή, ο συνάδελφο Κριστόφ Γουγιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βασικό θέμα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα είναι γιατί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, γιατί χρειαζόμαστε προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, διότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι σαν ε, τη, Σαν τη μαγιά για το Έχουμε 1,3 ευρώ που δώσαμε την πολιτική συνοχή για να μειώσουμε τι ε, διαφορέ μεταξύ των περιφερειών και να δώσουμε για την κοινή ευημερία των κρατών. Όμω σήμερα χρειάζεται να πολεμήσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε επιδοτήσει για τι περιοχέ μα, γιατί η Ευρώπη είναι παντού σε γονεί του δρόμου. Η πολιτική συνοχή έχει αλλάξει προ το καλό την εικόνα, το πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και επειδή χρειαζόμαστε να υποστηρίξουμε τι επιχειρήσει μα, διότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη υποστήριξη καινοτομία. Κύριε Αρτουή, έχω μια ερώτηση να σα θέσω. Είμαστε γείτονε, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ε, από γειτονικέ περιοχέ η Ευρώπη συνέβαλε πολύ για τη μικρή γεωργία, μικρή κλίμακα γεωργία. Χρησιμοποιήσουμε καλά του πόρου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Χρειάζεται μια απλούστευση ε, και ποια είναι τα μέσα τα οποία θα οδηγήσουν στην απλούστευση. Δεύτερον, πώ μπορούμε να γνωστοποιήσουμε καλύτερα τι πολιτικέ τη Ένωση και εκεί έχουμε μεγάλη προσπάθεια που να καταβάλουμε όσον αφορά την επικοινωνία. Πώ μπορούμε στον επόμενο προπολογισμό να έχουμε τα μέσα ούτω ώστε να εφαρμόσουμε την πολιτική επικοινωνία και να προσεγγίσουμε τους ε, πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο του ώστε να μπορέσει να απαντήσει στα διάφορα θέματα που εφήγησαν στι ερωτήσεις σας και στις προτάσεις σας. Πόσο χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε? Μέχρι τις 18.30 έχουμε στη διάθεσή μα. Αλλά εσεί μπορείτε να μείνετε εδώ αν θέλετε. Καλώ. Μάλιστα. Πάντως ε, πρόσεχω ιδιαίτερος στις παρατηρήσεις σας και διαπιστώνω σε τι βαθμό η πολιτική συνοχής είναι νευραλγική σημασία. Είναι σαν τις, ε, είναι μια αγελάδα μαζί με την κοινή γεωρική πολιτική. Ο κ. Χάσμαν μίλησε για την ανάγκη καλής συνεργασίας και της διαφύλαξης της πολιτικής συνοχής στα τωρινά επίπεδα. Έχουμε ένα νέο μηχανισμό, το InvestEU, όταν ο πρόεδρο Γκουνκέρα ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Νοεμβρίου του 2014. Έκανε τη διάγνωση ότι από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέφερε από ένα έλλειμμα επενδυτικό. Και μάλιστα ε, διαπίστωσε ότι στο τότε τότε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είχε αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά του. Οπότε όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα ε, η λύση είναι η μόχλευση και έτσι επινόησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και ορίσαμε έτσι τους κανόνες ώστε να μπορούν όλες οι περιφέρειες και όλες οι χώρες να υποφεληθούν από αυτό το εύση. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που διαχειρίστηκε πολλά κονδύλια μου είπε ότι όντω υπήρξε μια ακριβωδίκαιη κατανομή πέραν των αμυγώσεων δημοσιονομικών μέσων με τη μορφή επιδοτήσεων ή ενισχύσεων. Είχαμε ακριβωδίκαιη κατανομή. Βέβαια, μερικέ ε, ε, λύσει δόθηκαν χάρη ε, στο πρώην ΕΦΣΥ που τώρα ονομάζεται InvestEU. Είναι όμως το ίδιο όργανο που ουσιαστικά έχει συγχωνεύσει προηγούμενα ταμεία με επιπλέον στοιχείο την ελαστικότητα. Γιατί στο παρελθόν όταν ε, στέρευε ένα ταμείο περνούσαμε σε άλλο και με αυτές τις μεταφορές χάναμε χρόνο. Οπότε να έχετε κατά νου στις ε, πολιτικές σας, τις περιφερειακές, ότι χάρη στο InvestEU κάποιες επενδύσεις που δεν είχαν, ληφθεί, που δεν είχαν αναλυθεί από την αγορά μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, γιατί πια δίνεται, επένδυση, δίνεται εγγύηση από το πρόγραμμα InvestEU. Η κυρία Ταμάρα μας είπε ότι 4 στους 5 πολίτες ε, μένει, στο μέλλον θα μένει, 4 ε, στους 5 πολίτες θα μένουν στις πόλεις. Και επίσης είπατε ότι στηρίζετε τους προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση των αστικών κέντρων των πόλων και σίγουρα αυτή τη λίστα πρέπει να την διερευνήσουμε και να την στηρίξουμε. Και στο μέλλον να έχουμε ε, αρκετά ελαστικές διατάξεις ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές όταν ε, χρειάζεται να προσφύγουμε σε τέτοια κονδύλια, σε τέτοιες πιστώσεις. Ο κ. Κραβέκ είπε θα ήθελε η πολιτική συνοχή να γίνει το μέσο της αλληλεγγύης, να γίνει το εργαλείο της ελεγγύης, ώστε οι χώρες που δεν είναι κατάλληλα φορτιασμένες και εξοπλισμένες να καλύψουν το χαμένο έδαφος με τις πιο προηγμένες. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία. επίσης είπατε ότι οι μελλοντικέ επενδύσει θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παιδεία και την κατάρτιση. Όχι μόνο στις υποδομές στο κατασκευαστικό κλάδο. Είναι καλή η επένδυση για το μέλλον, η επένδυση στην παιδεία και στην κατάρτιση και σίγουρα δεν ε, ε, αμφισβητούμε που δεν είναι την αρχή της επικουρικότητας. Ο κύριος Φλεγκό μίλησε για την ασφάλεια και την ανάπτυξη και επέμεινε στην ανάγκη να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα θέματα της εκπαίδευσης. Επίσης, αυτά που είπε για τις ε, προσδοκίες της κοινωνίας και το κλίμα ε, σίγουρα η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτό το προβληματισμό της κοινωνίας το, για το κλίμα, για την υγεία, για το περιβάλλον. Και πιστεύω ότι η Ευρώπη που θέλει να επανασυμφιλιώσει αυτό το κενό και την ασυνενωσία που υπάρχει μεταξύ του γεωργικού κόσμου και των προστοκιών της κοινωνίας είναι να εφαρμόσει τις ίδιες διατάξεις παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα πάρει τις παρεξηγήσεις. Και στην εμπορική μας πολιτική, όταν συνάπτουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και αυστηροί, θα πρέπει να επιβάλλουμε στις ε, χώρες που εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλλουμε στις χώρες αυτές τις ίδιες συνθήκες παραγωγής και τους ίδιους όρους παραγωγής. Μόνο έτσι θα έχουμε ουσιαστικό αντίκτυπο και θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά το κλίμα. Ο κ. Να μίλησε για την ευθύνη των κρατών μελών και για τις συνέπειες του Brexit. Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, ίσως κάποιους μήνες μέχρι ότου διαλευκανθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, είμαστε στην ίδια γραμμή πλεύσης. Ε, και ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι μία από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, οι αντιδράσει του Συμβουλίου μέχρι στιγμής δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικέ. Και εδώ είναι θέμα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Ε, ό,τι αφορά τη φορολογία μπορεί μόνο με τα απομοφωνία να εγκριθεί και εκεί ανακύπτουν κάποια παζαρέματα και δοσοληψίες. Κύριε Τουρκ, μιλήσατε για την βιώσιμη αστική πολιτική και τα μέσα που θα τις αφιερώσουμε. Και Επισημάνεται και άλλες προκλήσεις όπως την ψηφιοποίηση. Ο κύριος Κάιζερ είπε ότι ο προϋπολογισμός καθορίζει την πολιτική. Αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και αντίστροφα. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τι πολιτική θέλουμε να επιδιώξουμε και μετά να αναζητήσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να την υλοποιήσουμε. Φυσικά λαμβάνοντα υπόψη το ρόλο και των περιφερειών και θα πρέπει να δείξουμε και θάρρος. Επιμείνατε στους φόρους, στη φορολογία, αλλά και εκεί αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη φορολογία και να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείξους, τις ε, παραδείξεις, τις φορολογικές απάτες, τη φοροδιαφυγή, τον ε, θετικό φορολογικό σχεδιασμό, μόνο η Ευρώπη θα μπορεί να εξασφαλίσει τα μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα προς τους πολίτες. Ε, με σεβασμό φυσικά και της διαφορετικότητας των περιοχών. Ο κύριος Μπόκ μίλησε για τις επενδύσει στην νεολαία, τον πολιτισμό, τη συνοχή και την ανάγκη να δώσουμε ψυχή, να εμφυσίσουμε πνοή στην πολιτική, στην ευρωπαϊκή πολιτική και να ορίσουμε σωστά τους στόχου της πολιτικής. Και αν αυτή τη στιγμή ε, οι συνθήκες δεν προβλέπουν κοινοτική αρμοδιότητα για την παιδεία, ούτε για την επαγγελματική κατάρτιση, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ε, για να προχωρήσουμε και το Έρασμος είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Το 2017 είχαμε την 30η επέτειο του Έρασμος, αλλά θα πρέπει να εκδημοκρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί προς το παρόν το έρασμο εξυπηρετεί κυρίω φοιτητέ ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημίων. Δεν μπορούμε όμω να αφήσουμε άνεργου νέου ή ε, νέου που έχουν εγκαταλείψει τι σπουδέ. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και για αυτού, να βοηθήσουμε και αυτού του νέου. Και το ενδιαφέρον της κινητικότητας είναι ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν επιτύχει περισσότερο από εμά και να τους εμφυσίσουμε ή να τους εμπνεύσουμε με καλές πρακτικές. Κύριε Ντρομπρά, κυρία Ντρομπρά, δεν θυμάμαι πια. Ζητώ συγγνώμη, αναφέρθηκε στην πρόκληση της ασφάλειας, στην πολιτική συνοχής και την ανάγκη για ευελιξία. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατο σημείο. Ε, Ξεπλάγινα από τη σημασία του δημοσιονομικού μας κανονισμού. 500 ε, σελίδες αποτελείται. Σαν υπήρχε κακά, καχυποψία όσον αφορά τη σύλληψη του κανονισμού. Δεν κάνουμε τίποτα με την καχυποψία. Αν φαίνεται ότι κάποια κράτη έχουν προβλήματα, δυσκολίες να ασκήσουν το δημοσιονομικό έλεγχο ικανοποιητικά. Ίσως θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τι χώρες συγκεκριμένα. Αυτός δεν είναι όμως λόγος, δικαιολογία. Διότι κάποιες χώρες έχουν σύστημα ε, δημοσιονομικού ε, ε, ελέγχου που είναι κάπως απερχιωμένο να επιβάλλουν κανόνες και σε χώρες που έχουν τα καλύτερα μέσα ελέγχου. Δεν θα πρέπει να διστάζουμε να θεσπίζουμε την ευελιξία. Δεν μπορούμε να, να έχουμε στενούς κανόνες και να τονίζουμε ότι χρειάζεται καινοτομία. Αν έχουμε απειρχιωμένους κανόνες σε ένα θεσμό στην Ευρώπη που δεν έχει κυβέρνηση αλλά έχει ε, νομική βάση και κανόνες ίσως να έχουν συγγραφεί κάποιοι κανόνες μια εποχή που τα προβλήματα που πρέπει να διφετήσουμε τώρα δεν είναι τίθεντο. Είναι παλιοί κανόνες. Εξού και η δυσκολία όσον αφορά τη μετανάστευση όσον αφορά τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης, όλα αυτά άλλαξαν τα δεδομένα και κάποιες βάσεις πρέπει να αναθωρηθούν. Και νομίζω έχουμε λόγο να επιμένουμε επί της αναγκαίας ευελιξίας. Κύριε Ρουγιό, όπως και εσείς είμαστε από κοντινή περιοχή, ανήκαμε στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια επαρχία, γιατί ο ίδιος προπολογισμό για να εφαρμόσουμε μια πολιτική, καλό θα ήταν να διεξαχθεί μια συζήτηση πιο καλά διαρθρωμένη, λεπτομερέστερη όσον αφορά το τι προτιθέμεθα να κάνουμε με την Ευρώπη πριν αποφασίσουμε τον προπολογισμό. Έτσι που έχει ετοιμαστεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν λέω ότι είναι business as usual, αλλά κάπως ε, αλλάζουμε ε, την κατάσταση χωρίς να θέτουμε το θεμελιώδες ερώτημα. Δεν θέλουν να χαλαρώσουν τα κράτη-μέλη. Κατάλαβα ότι η τοπική αυτοδίκηση και εγώ σαν ερετός εκπρόσωπος τοπικής αυτοδίκησης που είμαι, έχω ζήσει σε αυτό το τομέα είναι καλύτερο υπάρχει εμπιστοσύνη και απλούστευση, καλύτερη επικοινωνία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι θέλουμε για επικοινωνία αλλά θα πρέπει να έχεις κάτι να πεις άμα έχεις την επικοινωνία για να επικοινωνήσεις από καιρού καιρών λοιπόν θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις που να ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη Τούτου λεχθέντος σας λέω ότι καρπός των εργασιών της Επιτροπής σας είναι η αυτοπεποίθηση που με διακατέχει και η εμπιστοσύνη με διακατέχει. Θα πρέπει να συντονιστούμε, να κινηθούμε προς όφελος Ευρώπης, να την κάνουμε παγκόσμια δύναμη που θα προετοιμάσει το μέλλον μας και που θα μας προστατεύει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτήν την τόσο έντονη συζήτηση όπου συμμετείχαν τόσο πολλοί συνάδελφοι από την Επιτροπή μας. Αυτό ήταν ο στόχος. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, να δούμε τι συνέχεια δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις μας. Σε τρεις ολομέλειες εργαστήκαμε πολύ για τις γνωμοδοτήσεις αυτές. Ακούσαμε σήμερα πώς έχουν τα πράγματα σε αυτήν την ενδιάμεση φάση. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί αποδεικνύει ότι αυτά που κάνουμε εδώ σε κάτι χρησιμεύουν. Και τώρα θα ξεκινήσει το τελικό sprint για να νικήσουμε αφού θα καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας ε, το Συμβούλιο Υπουργών. Ευχαριστώ, διακόπτουμε μέχρι αύριο σε 9. Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, για την παρουσία σας και σας εύχομαι μια ευχάριστη βραδιά.